Buongiorno a tutti. Cominciamo che sono le 9.05. E Καλημέρα. Ξεκινάμε σε 9 και 5. Innanzitutto Λοιπόν, πρώτα απ' όλα χαιρετίζουμε νέο υπάλληλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Κρίστοφ Μέρλικ, του ευχόμαστε καλή δουλειά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως πάντα, απευθύνεται μέσω web streaming η συνεδρίασή μας και έχει διαβιβαστεί διόντως και ημερήσια διάταξη. Το πρώτο σημείο της ημερήσια διάταξης είναι η απαλλαγή του Κοινοβουλίου του 2009. Είναι εδώ εισηγητής ο συνάδελφος Ιταλά, στον οποίο δίνω το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Καταφέραμε να συνεργαστούμε άριστα όσον αφορά το σχέδιο εκθέσεως. Η έκθεση συνετάχθη με τέτοιο τρόπο που οι επικεφαλεί των μονάδων εξέτασαν τα ζητήματα, συζητήσαμε με πολλούς υπαλλήλου τα θέματα αυτά και εξηματούχους. Το 2009 ήταν ιδιαίτερο έτος από πολλές πλευρές. Διεξήξαν εκλογέ, βέβαια και επιπλέον είχαμε και το νέο καταστατικό για τα μέλη και για τους βοηθούς και τα νέα αυτά καταστατικά δημιούργησαν προβλήματα όσον αφορά την αρχική εφαρμογή των αποφάσεων. Δημιουργήθηκε μια επιτροπή ad hoc η οποία εξέτασε τα δύσκολα θέματα, προσπάθησε να βρει λύση και θα έλεγα ότι είμαστε σε καλύτερη θέση τώρα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι τα νέα καταστατικά για τα μέλη είναι το νέο καταστατικό για τα μέλη είναι τέτοιο που προβλέπει μια νέα υπηρεσία για τα μέλη και υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Πιστεύω ότι η κατάσταση είναι καταστροφική όσον αφορά την έλλειψη προσωπικού. Δεν υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να γίνει και θα έλεγα ότι ότι δεν προετοιμάστηκαν με διεξοδική ανάλυση τα νέα καταστατικά. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα-δύο θέματα, θέματα τα οποία θα ήθελα να υπογραμμίσω, θέματα της εκθέσεως. Κάτι πολύ επίκαιρο είναι η ασφάλεια. Το 2008 κάναμε μία πρόταση όσον αφορά τη βελτίωση ε, την ασφάλεια χρησιμοποίησαμε όλο και περισσότερα χρήματα για την ασφάλεια, τη σωματική ασφάλεια και την ασφάλεια από πλευρά επιθέσεων. Βάλαμε περισσότερους φρουρού, κάμερε. Παρ' όλα αυτά έγινε μια ληστεία τράπεζας και την περασμένη Παρασκευή μάλιστα έγινε και ληστεία στο ταχυδρομείο. Και κανεί από τους ε, ενόχους δεν ε, συνελήφθη. Βέβαια απ' έξω γελούν μαζί μας. Τι είδους ασφάλεια έχουμε εδώ μέσα. Και βέβαια τα μέλη μπορούν να κοιταχθούν στον καθρέφτη διερωτώμενοι για το θέμα, διότι τα μέλη πήραν τις αποφάσεις όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα μέλη να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική αυτή ταυτότητα, το badge, για να μπουν στο κτίριο. Τα μέλη μπορούν να περπατούν εντός του κτιρίου ελεύθερα και υποτίθεται πάντα ότι οι φρουροί πρέπει να ξέρουν και τους 736 βουλευτές. Ξέρουμε ότι αυτό είναι αδύνατον. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιοι μπαίνουν από το δρόμο, περνάνε από το διάδρομο των ευρωβουλευτών, λένε καλημέρα στους φρουρούς, σαν να είναι ευρωβουλευτές, και παίρνουν το δρόμο τους. Ε, δόθηκε πολύ μεγάλη δημοσιότητα στη ληστεία, στις ληστείες που έγιναν εδώ και πόσο εύκολο είναι να δυσδύσει κανείς να εισχωρήσει στο κτίριο και θα ξέρουν και οι τρομοκράτες ότι είναι εύκολο στόχος. Άρα πρέπει να βελτιώσουμε την, τα μέτρα ασφαλείας. Ε, δεν καταλαβαίνω την αρχή αυτή που ακολουθείτε. Δηλαδή ότι οι βουλευτές δεν είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό τους αυτό badge, το ηλεκτρονική, την ηλεκτρονική ταυτότητα και κάποιοι μπαίνουν μάλιστα και ξαναβγαίνουν αμέσως α, χωρίς να υπάρξει ο παραμικρός έλεγχος. Αν πιάσει φωτιά το κτίριο, κανείς δεν θα ξέρει ποιοι ευρωβουλευτές είναι στο κτίριο και ποιους πρέπει να ψάξουμε αν πιάσει φωτιά. Huonosti hoidettu ja selvästi muutos. Νομίζω ότι δεν υπάρχει σωστή αντιμετώπιση. Πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Όσον αφορά τη διαδικασία υπογραφής, ο, α, υπογράφουμε, βάζουμε την υπογραφή μας την Παρασκευή όταν δεν υπάρχουν συνεδρία. Πρέπει να υπογράψουμε. Και έμεινα έκπληκτος διότι πολλοί υπάλληλοι που ασχολούνται καθημερινά με αυτά τα θέματα εξετάζουν τις υπογραφές και εισάγουν στη βάση δεδομένων όλα τα ονόματα τη υπογραφέ. Τεράστιο φόρτος εργασία. Αν μπορούσαμε χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική μας ταυτότητα, όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν ηλεκτρονικά και θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε πολλά χρήματα, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να εξοικονομήσουμε χρόνο. Και θα ήταν κάτι καλό και από πλευρά ασφαλεία. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποιε αλλαγέ. Και είναι δύσκολο να συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε το παρόν σύστημα. Όσον αφορά τις κάμερες, ε, την περασμένη Παρασκευή λοιπόν, όπως σας είπα, έγινε μια ληστεία στο ταχυδρομείο και πράγματι διαπιστώσαμε ότι λειτουργούν οι κάμερες και είχαμε εικόνες των ε, ληστών. Είμαι σίγουρος ότι το γεγονός ότι είχαμε κάμερες στο κτίριο ήταν κάτι που μας επέτρεψε να έχουμε εικόνες αυτών των εγκληματιών και ελπίζω ότι αυτή η συγκεκριμένη υπόθεση θα καταλήξει αίσια όσον αφορά το, την ανακάλυψη και σύλληψη των ληστών. Πηγαίνοντας πίσω δύο Παρασκευές, ήμουνα στο κτίριο όταν ληστεύτηκε το αχυδρομείο. Ε, Έφερα από το κτίριο λοιπόν και κανείς δεν ε, μπορούσε να βγει από το κτίριο, δεν το επιτρεπόταν. Και εγώ ρώτησα ποιο θα μου πληρώσει το νέο μου εισιτήριο το αεροπορικό, διότι δεν με αφήναν να φύγω από το κτίριο. Και όταν ρώτησα το φρουρό, τους φρουρούς, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω, μου λέει ο φρουρός, για λόγους ασφαλείας. Τι ασφαλείας του λέω. Και μου λέω, κοίτα να δεις, φεύγει η πτήση μου, πρέπει να βγω από το κτίριο. Θα μ' άρεσε, θα ήθελα όλοι οι βουλευτές να ήταν εδώ και να βιαζόταν όλοι οι βουλευτέ να πάνε κάπου και οι φρουροί να λένε Συγγνώμη, δεν πάτε πουθενά για λόγου ασφαλεία. Είμαι σίγουρο ότι αν αυτό είχε συμβεί, θα χτυπάγαμε τα πόδια μα στο πάτωμα και θα πετούσαμε αλλαγή των μέτρων ασφαλεία. Δεν μα άφησαν να φύγουμε, δεν μα είπαν καν πότε θα μα επιτραπεί να φύγουμε και κανεί δεν ήξερε αν θα καταφέρει να προλάβει την πτήση του. πάντα στο θέμα της ασφαλείας και της συνεργασίας με την αστυνομία. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε πολύ καλύτερη συνεργασία με την αστυνομία. Κάποτε ε, παρκάρισα το αυτοκίνητό μου στη Ρίου γιατί βιαζόμουν να πάω στη συνεδρίαση. Μετά από μισή ώρα πάω να πάρω το αυτοκίνητό μου και τα λάστιχά μου τα είχαν κομματιάσει. Και όταν ζήτησα βοήθεια από τους φρουρούς για να μου πούν τι συνέβη, οι φλουροί μου λένε λυπάμαι, εμείς δεν ανακατευόμαστε. Και η αστυνομία είπε συγγνώμη, είμαστε ομοσπονδιακή αστυνομία και όχι αστυνομία των Βρυξελών, δεν μπορούμε με το θέμα. Καμιά φορά φαίνεται ότι δεν υπάρχει παραμικρή συνεργασία με την τοπική αστυνομία. Τώρα πάω σε άλλα θέματα και πιο συγκεκριμένα το προσωπικό του Κοινοβουλίου και η ανάθεση σε εξωτερικούς φορείς διαφορών εργασιών. Ε, είχαμε αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες πάρα πολλές δραστηριότητε, κυρίως στην τεχνολογία της πληροφορικής. Είχαμε πάρα πολλά προβλήματα και έπρεπε να, πρέπει να προσέξουμε μάλλον πάρα πολύ την πολιτική που ακολουθούν σε αυτόν τον τομέα. Διότι αν αναθέτεις έξω τα πάντα, ε, τελικά θα είναι αυτή η λύση πάρα πολύ δαπανηρή. Άρα υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης για πιο πρακτικά ζητήματα τώρα. Υποτίθεται ότι θα ήταν έτοιμο ένα κέντρο επισκεπτών και θα ήταν έτοιμο μέχρι το 2009 και ακόμα δεν είναι έτοιμο. Και οι λόγοι για τους οποίους δεν είναι έτοιμο το κέντρο επισκεπτών ε, δεν ακούγονται πολύ πιστικοί. Κάποιος είπε ότι ο χώρος ήταν εγκαράς πριν και γι' αυτό το λόγο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει το χτίριο. Όλοι το ήξεραν όμως από πριν, όταν είχαν καθορίσει την ημερομηνία. Άρα υπάρχουν κάποια εκκρεμή ζητήματα όσον αφορά το θέμα και τα ηλικιωμένα άτομα όταν θέλουν να πάνε, στην, να πάνε στα θεωρία για να παρακολουθήσουν την Ολομέλεια πρέπει να περάσουν επανειλημμένα από σημεία ασφαλείας Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερο σχεδιασμός για τους επισκέπτες. Και βέβαια πρέπει να δούμε και τι θα κάνουμε με το κέντρο των επισκεπτών. Η ο... Όσον αφορά τις ομάδες επισκεπτών, η ομάδα ελέγχου είπε ότι όταν έρχονται εδώ επισκέπτες, πολύ συχνά πληρώνουν σε ρευστό διοικητικές δαπάνες. και καταβάλλεται ένα καταποκοπήν ποσό ανεξάρτητα από τις πραγματικές δαπάνες. Κάποιοι τελικά φεύγουν με λεφτά στο χέρι και κάποιοι μένουν χωρίς χρήματα για την επίσκεψή τους, διότι εξαρτάται από πού ήρθαν αυτοί οι επισκέπτες. Πρέπει να το εξετάσουμε, πρέπει να δούμε ποια είναι η πραγματική δαπάνη για τους επισκέπτες και θα πρέπει να αποζημιώνουμε για το πραγματικό κόστος, βέβαια σε κάποια όρια, ε, διότι δεν μπορούν να μένουν όλοι στο Χίλτον και να τρώνε σε εστιατόρια του καταλόγου Μισελά. Ε, θα πρέπει να βλέπουμε ποια είναι, ποιο είναι το πραγματικό κόστος. Έχουμε τη δική μας τηλεόραση του διαδικτύου, Web TV, και βλέποντας πόση προσπάθεια καταβάλει στον τομέα, πόσα χρήματα δίνουμε και πόσοι είναι οι θεατές, δεν νομίζω ότι τελικά αυτή η επένδυση ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν είμαι καν σίγουρος κατά πόσο η αρχή ε, ύπαρξης δικού μας ε, καναλιού δικαιολογείται. Υπάρχει, υπάρχουν ελεύθερα μέσα ενημέρωσης και αναφέρουν αυτά που κάνουμε εδώ δεν είμαι σίγουρο ότι χρειαζόμαστε τη δική μας τηλεόραση, τη δική μας web TV. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν πάρα, δεν ήταν πάρα πολύ επιτυχής. Αν δείτε τα αποτελέσματα, σχέση με τα ποσά που καταβάλουμε, δεν ήταν θετικά τα αποτελέσματα. Πέρσι μιλήσαμε για τα βραβεία και τα βραβεία για τους δημοσιογράφους. Είναι λίγο παράξενο το ότι τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να επικρίνουν πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά δίνουμε και βραβεία σε δημοσιογράφου που ήταν οι καλύτεροι και οι πιο ευγενικοί σε εμά. Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι αυτό είναι πάρα πολύ δημοκρατικό. Δεν είμαι σίγουρο ότι είναι καλή χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων αυτά τα βραβεία. Ίσως θα έπρεπε να εστιαστούμε επί των βασικών μα καθηκόντων ανταυτού. Μετά, όσον αφορά τη διερμηνία, Υπάρχουν πολλά προβλήματα που σχετίζονται με αυτό το θέμα. Θα πρέπει να προσέξουμε βέβαια ότι στο μέλλον θα έχουμε προβλήματα αν 15 κράτη-μέλη, οι διερμηνείς 15 κρατών μελών συνταξιοδοτηθούν. Θα υπάρξει εκεί ένα πρόβλημα, πρόβλημα γενεών και δεν έγιναν αρκετά πράγματα για να υπάρχει σωστό ρυθμό αντικατάσταση εκείνων που βγαίνουν σε σύνταξη και αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε αρκετού μεταφραστέ ή διαρμηνεί στο μέλλον. Άρα πρέπει να είμαστε σε καλύτερη επαφή με τα κράτη-μέλη, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι το σύστημα θα διοργανωθεί με το βέλτιστο τρόπο. Όσον αφορά το ταξιδιωτικό γραφείο, υπήρξαν πολλά προβλήματα και με το ταξιδιωτικό γραφείο. Αν δείτε ένα γραφείο ταξιδίων που έχει το μονοπόλιο της διοργάνωση των ταξιδίων μας. Και τελικά αυτό το εξαιρετικό γραφείο οδήγησε πολλούς ευρωβουλευτές να πάνε στο διαδίκτυο να δούνε ποια είναι η τιμή του εισιτηρίου κοιτάνε και αντιμέτωπη του εισιτηρίου οι βουλευτέ στο διαδίκτυο και όταν πάω στο ταξιδιωτικό γραφείο το ίδιο εισιτήριο είναι δύο-τρει φορέ ε, πιο ακριβό. Γιατί ξέρει το ταξιδιωτικό γραφείο ποιο είναι το ανώτατο όριο και βάζει την τιμή στο ανώτατο όριο. Ε, δεν νομίζω ότι αυτή είναι η καλή, καλή προσέγγιση όσον αφορά τη χρήση των χρημάτων του φορολογουμένου. Μετά άλλο θέμα. Ερώτηση. Τι γίνεται όταν αλλάζουμε ταξιδιωτικό γραφείο. Είχα ένα ταξιδιωτικό γραφείο που είχε εκδώσει ένα εισιτήριο, αλλά αυτό το εισιτήριο δεν ίσχυε πια όταν πήγα στο αεροδρόμιο. Το ταξιδιωτικό γραφείο είχε κάνει λάθος, αλλά δεν με αποζημίωσαν αμέσως. Μου ζήτησαν να γεμίσω διάφορες σελίδες, να έρθω την επόμενη εβδομάδα και μετά την άλλη εβδομάδα και τελικά μου είπαν «Ούψ, λυπάμαι, αυτό ήταν το παλιό γραφείο ταξιδιωτικό που εξέδωσε το, το εισιτήριο και το νέο ταξιδιωτικό γραφείο δεν είναι υπεύθυνο για αυτά που έκανε το παλιό ταξιδιωτικό γραφείο, άρα την πατήσατε». Φαίνεται λοιπόν ότι όταν αλλάζουν τα ταξιδιωτικά γραφεία, φεύγει το ταξιδιωτικό γραφείο, μένουν πίσω και παίρνουν μαζί τους, αφήνουν τις αφήνες τους, δεν τις αναλαμβάνουν. Όσον αφορά το μηχανισμό εθελοντικής συνταξιοδότησης, μας μίλησαν οι για αυτό το θέμα και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τελικά θα πρέπει να ανταποκριθεί στις καταστατικές του ευθύνες του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τις συνταξιδοτήσεις. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την κατάσταση διαφορετικά. Θα καταλήξουμε σε παράλογη κατάσταση. Θα έχουν ε, βουλευτέ βάλει χρήματα σε συνταξιωτικό ταμείο και δεν θα μπορέσουν να πάρουν τα χρήματά του να βγουν στη σύνταξη. Και αυτό δεν είναι νόμιμο. Και Πρόεδρε, κάποια άλλα ίσον σημασία θέματα. Πολύ συχνά μιλάμε για το γεγονός ότι τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές θα πρέπει να είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Συνεχώς παράγουμε νομοθεσία που επιβάλλεται στους απλούς πολίτες, επιβάλλουμε περιορισμούς αυτούς, αλλά δεν επιβάλλουμε περιορισμούς στους αυτούς μας. Δεν το κάνουμε αυτό όταν δούμε τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούμε για την μεταφορά μας. Νομίζω θα πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις για να είμαστε πιο περιβαλλοντικά φιλικοί και να συμμορφωθούμε καλύτερα με τις νομοθεσίες μας. Κάποιοι βουλευτές που έρχονται εδώ με τα παιδιά τους, και βάζουν τα παιδιά τους στο ευρωπαϊκό σχολείο. Εδώ υπάρχει κόστος μεταφοράς πέραν των 2.000 ευρώ το χρόνο. Τώρα, είναι αρκετά αυτά τα πόσα ε, μιλήσαμε στην Κομισιόν γι' αυτό και ήταν το Συμβούλιο που είχε αποφασίσει το θέμα αυτό στην πραγματικότητα και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνεται διάκριση κατά του Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό, διότι όλοι οι άλλοι έχουν αυτό το, ε, το ωφέλιμα. Είτε όλοι θα πληρώνουν, είτε κανείς. Ε, δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Υπάρχει μια διαφήμιση έξω που λέει ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να συμφιολιώσει την εργάσιμη ζωή με την οικογενειακή ζωή. Και όταν φέρνει ε, ο βουλευτής την οικογένειά του εδώ, έχει να καλύψει αυτά τα έξοδα μεταφοράς των παιδιών στο σχολείο. Δεν είναι σωστό αυτό. Θα πρέπει να έχουμε και εμείς την ε, ελευθερία επιλογή στο θέμα αυτό. Ένα άλλο πιο δύσκολο, πιο ευαίσθητο θέμα τώρα έχουμε τις τρει έδρε. Βρυξέλλες, Στρασβούργο, Λουξεμβούργο. Δεν θα τοποθετηθώ ως προς το πού πρέπει να είμαστε, γιατί η απάντηση θα είναι το Στρασβούργο. Αλλά ε, Είμαστε σε αυτή την οικονομική κατάσταση που είναι δυσχερής και ε, γνωρίζω ότι το Συμβούλιο θα ζητήσει από το Κοινοβούλιο να κάνει περικοπές δαπανών απαντησα θα πρέπει να πούμε στο Συμβούλιο ότι Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να ε, κάνουμε εξοικονομήσεις 200.000 ε, ε, ευρώ το, το χρόνο. Να, γίνεται, να υπάρχει μόνο μία έδρα. Αλλά ο κόσμος δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να είμαστε σε τρει έδρε. Και εμεί λέμε αυτό ε, υπάρχει στη συνθήκη. Αλλά η συνθήκη έχει τροποποιηθεί προς το καλύτερο σε πολλά σημεία. Και δεν κατανοώ γιατί δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε τη συνθήκη έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε ε, κονδύλια και να μην χρειάζεται κάθε τρεις εβδομάδες να πηγαίνουμε σε άλλες ε, τοποθεσίες. Πρέπει να εξοικονομήσουμε χρήματα και ξέρει το Κοινοβούλιο πού μπορεί να εξοικονομηθούν αυτά τα χρήματα. Ευχαριστώ κύριε Ήτελα. Ας περάσουμε στη συζήτηση. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή ε, για τα όσα είπε και για την προσήλωσή του ε, στην υπόθεση αυτή της απαλλαγής του Κοινοβούλιο το 2009. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την εξής γενική παρατήρηση. Η ομάδα μου φρονεί ότι θα πρέπει να είμαστε όσο γίνεται πιο διαφανείς για το δικό μας προπολογισμό και για την ευθύνη που φέρουμε. Αυτό δεν το λέω μόνο λόγω της σημασίας του Κοινοβουλίου αυτής καθ' αυτής, και, αλλά ε, και για τη σχέση μας με το Συμβούλιο. Γιατί έχουμε ενισχύει αυτή την περίεργη συμφωνία κυρίων που καλό θα ήταν κατά μένα σιγά σιγά να την καταργούμε. Θα πρέπει ο καθένα να φροντίζει για πλήρη διαφάνεια. Και η ομάδα μου θεωρεί ε, ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν ε, με τρόπο λογικό και φρόνιμο και ως ενήλικες να αρχίσουν να συζητούν και τέτοια πράγματα. Έρχομαι στην ουσία τώρα. Υπάρχουν μερικά θέματα που θα ήθελα να τα αναφέρω αλλά με κάλυψε και ο εισηγητής σε αυτά, τα ανέφερε και ο ίδιος. Το πρώτο είναι η χρήση του χαρτιού στο κοινοβούλιο. Το 2009 πετάξαμε χίλιους τόνους χαρτί. Ε, δεν το πετάξαμε ακριβώς. Υποτίθεται ότι ανακυκλώνεται στη συνέχεια αλλά είναι τεράστια κατανάλωση χάρτου εδώ στο Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι επεξεργάζονται ορισμένοι κάποια συστήματα για να χρησιμοποιούμε περισσότερο τις ηλεκτρονικές μορφές επικοινωνίας. Ε, η ε, πολιτική μου ομάδα θέλει να επιταχυνθεί αυτή η προσπάθεια. Θεωρώ άχρηστο σε κάθε συνεδρίαση που ερχόμαστε να έχουμε όλα τα έγγραφα ένα έτοιμα. Έχει προχωρήσει πια η τεχνολογία αρκετά, ώστε να έχουμε πολύ πιο εύκολα συστήματα έχει το καθένας με το iPad, με τον υπολογιστή του. Δεν χρειάζεται να τα έχει όλα τυπωμένα. Εξού και οι χίλιοι μπορούν να μειωθούν. Το σύρματο διαδίκτυο θα πρέπει να επιταχυνθεί και γρήγορα να βελτιωθεί, αλλά έχω καταλάβει ότι και με αυτό ασχολούνται οι υπηρεσίε. Δεύτερον, η ασφάλεια. Συμφωνώ με τον εισηγητή, όσα είπε προηγουμένω. Εξεπλάγει αυτή την εβδομάδα για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται στους βουλευτές. Όλοι θέλουν να ενταθούν τα μέτρα ασφαλείας και διαπιστώνω και παρατηρώ ότι και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου μας ακόμα δεν θέλει να το εφαρμόσει αυτό. Να μπαίνουμε εμείς με την κάρτα εισόδου μας ως βουλευτές. Δεν καταλαβαίνω κι εγώ πως ο βουλευτής γιατί χωρίς να δίνουμε κανένα στοιχείο ταυτότητας να μπαίνουμε ωραία και καλά να παρελάβουμε από την είσοδο και όλοι οι υπόλοιποι να ανοίγουν με την ηλεκτρονική τους κάρτα τις πόρτες. Ε, αν η ασφάλεια επεκταθεί και στα μέλη του Κοινοβουλίου θα βελτιωθούν τα πράγματα. Δεν λέω ότι έτσι αποτραπούν οι ληστείες και επιθέσεις σε τράπεζες και ταχυδρομεία. Ε, αλλά α φροντίσουμε και οι βουλευτέ να βάλουμε και εμεί το λιθαράκι μα στην ασφάλεια. Τρίτο πρόεδρε. Τα κτίρια. Συμφωνώ με την κριτική του εισηγητή. Θα ήθελα να επαναλάβω κάτι η ρητά για το ευρωπαϊκό, οίκο ευρωπαϊκής ιστορίας. Έχει γίνει πια σύριαλ, σαπουνόπερα και σαπουνόπερα διαφανής. με πολύ αφρό. Δεν έχουμε δει ε, αρκετή πληροφόρηση ακόμα για αυτό το θέμα. Έχω επιχειρήματα να σας δώσω, αλλά κινδυνεύουμε να πέσουμε σε τεράστια καταστροφή και φιάσκο. Τι άλλα έχω εδώ, Πρόεδρε, που ήθελα να πω. Α, κάτι που έχει και πέρσι. Μετά το ψήφισμα, πέρσι, για την απαλλαγή. Παρακολούθησα την υπόθεση με τις υπηρεσίες. και πρέπει να σας πω για τα ποδήλατα στο Στρασβούργο. Ε, πώς έχει η κατάσταση. Είχα πει να αντικαταστήσουμε τα αυτοκίνητα, να αποσύρουμε ένα αυτοκίνητο και να βάλουμε δεν ξέρω πόσα ποδήλατα στη θέση του. Το Στρασβούργο προσφέρεται καταπληκτικά, είναι πάρα πολύ καλά εξοπλισμένο ως πόλη, ε, η πόλη του Στρασβούργου για ποδήλατα. Είμαι σε συνεννόηση με τι υπηρεσίε, Θυμάστε όλοι το σύριαλ, μάλιστα κύριε Υπουργέ. Yes, Minister. Ε, αυτό είναι ε, που συμβαίνει και εδώ στο Κοινοβούλιο. Τι θέλουν οι υπηρεσίες. Α, να μας διαθέσει, λέει, η πόλη του Στρασβούργου τα ποδήλατα, καμιά δεκαριά ποδήλατα για βουλευτέ και μόνο, αποκλειστικά. Εκατό χιλιάδε φορέ έχω πει ότι δεν θέλω να μου το διαθέσει ο Δήμος του Στρασβούργου, το Κοινοβούλιο ως θεσμό. Και αυτό έχει σημασία όχι μόνο για τα ποδήλατα αυτά καθ' αυτά και για την εικόνα που δίνουμε ότι ε, έχουμε και ποδήλατα, όχι μόνο κουρσάρες για τους βουλευτές. Και μπορούν οι βουλευτές να πάρουν το ποδήλατό τους και να κυκλοφορούν στο Στρασβούργο. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το επεισόδιο του Yes Minister. Ε, θα το συνεχίσω και αν δεν προλάβω να κάνω ε, κάτι μέχρι να ε, τελειώσουν οι προθεσμίες για τις τροπολογίες για την παρούσα έκθεση θα δω τι θα μπορέσω άλλο να κάνω. 100% τώρα, Πρόεδρε, των πτήσεων ε, που παίρνουμε για τη δουλειά μας θα πρέπει να το αντισταθμίζουμε το διοξίδιο του άνθρακα. Ακόμα δεν είναι αυτό γεγονός. Θέλω να επιταχυνθεί αυτό και ισχύει ε, και ε, το ίδιο με αυτό που είπα προηγουμένως. Θα κάνω τροπολογία εάν δεν βλέπω να προχωρούν γρήγορα τα πράγματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σόλτεβους. Tak Ευχαριστώ ε, τον κύριο Ιταλά για αυτή την έκθεση. Νομίζω περιέχει στοιχεία με τα οποία θα συμφωνούσα. Αυτό που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε σε αυτή την έκθεση είναι ένα κείμενο σχετικά με την οικονομική κρίση. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει περισσότερες εξοικονομήσεις και ε, στη χρήση κονδυλίων σε αυτή την περίοδο χρήσεως. Θα πρέπει να το θέσουμε και αυτό μέσα στην έκθεση. Αναμφίβολα υπάρχουν πολλά ε, παραδείγματα όπου αυτό δεν γίνεται. Για παράδειγμα, στα ταξίδια δεν έχει γίνει τίποτα. Όταν ε, ζητάμε ε, να μας διευθετήσουν ένα ταξίδι στο ταξιδιογραφείο δεν μας δίνουν πάντα την πιο ευνοϊκή προσφορά και, δεν, ε, και είναι το ταξιδιογραφείο το γραφείο που κερδίζει και αυτό δεν είναι λογικό. Γι' αυτό θα πρέπει να το γράψουμε αυτό στο κείμενο. Υπάρχουν πολλές καλές προτάσεις. Θα πρέπει να ενισχύσουμε, να διευκρινίσουμε ίσως ε, οι θέσει εργασίας μας ε, διακυβεύονται. Θα πρέπει να κάνουμε εξοικονομήσεις και γνωρίζω πολύ καλά ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν μπορεί να το αποφασίσει από μόνο του. Θα πρέπει να ζητήσουμε από τα μέλη να κάνουν αυτή τη συζήτηση με άλλα όργανα για τις εξοικονομήσεις. Μετά, το θέμα της ασφάλειας στο Κοινοβούλιο. Ε, είναι ένα πολύ επίκαιρο θέμα βέβαια αυτή τη βδομάδα, είναι ένα φλέγον θέμα. Ε, έχουμε ε, με μεγάλο αριθμό ατόμων που ασχολούνται με την ασφάλεια. Αυτή η δουλειά στον τομέα της ασφάλειας αναρωτιέται κανείς αν είναι αποτελεσματική όσο θα έπρεπε, αν είμαστε αποτελεσματικοί εμείς ήδη στην πολιτική ασφαλείας μας. Όλοι συμφωνούν ότι απαιτείται πολύς χρόνος στην καταχώρηση και την εγγραφή των επισκεπτών που στέκουν στην ουρά για να γραφτούν και αυτό δεν είναι αποδεχτό. Ε, πώς θα βελτιώσουμε την κατάσταση είναι το ερώτημα. Βεβαίως θα πρέπει να βρούμε λύσεις συμβιβαστικές. Συμφωνώ με τον εισηγητή που λέει ότι θα πρέπει να ρυθμιστεί και η πρόσβαση των βουλευτών. Θα πρέπει να συμβάλλουμε και εμείς στην ασφάλεια στο Κοινοβούλιο και θα πρέπει και εμείς να δεσμευτούμε να δείχνουμε την κογκάρδα μας, στην ηλεκτρονική ταυτότητα ή να ε, δεχτούμε μια ηλεκτρονική εγγραφή στο Κοινοβούλιο κανένα μέτρο δεν μπορεί να βελτιώσει την ασφάλεια όσο η δική μας θέληση. Η δική μας εγγραφή λοιπόν είναι απαραίτητη. Αυτό μας βοηθά να κάνουμε εξοικονομήσεις και να βελτιώσουμε και την ασφάλεια. Γενικώ ε, θα έλεγα ότι είναι μια καλή έκθεση. Έχω προετοιμάσει κάποιες τροπολογίες για να <clears throat> διευκρινιστεί η δική μας ε, οικονομική ε, υποχρέωση, για να κάνουμε πιο πράσινο το κοινοβούλιο και γενικά, επαναλαμβάνω, είναι μια καλή έκθεση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Herzog. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τους συζητητές και τον σκιωδή συζητητή και είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση κάθε χρόνο. Ε, ήμουνα πέρσι σκιώδης εισηγήτρια και ε, έχω μεγάλο ενδιαφέρον προς την βελτίωση της αποδοτικότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την οικονομική αποδοτικότητα αλλά και σε όλες τις διαδικασίες της. Ο λόγος που ζήτησα το λόγο και θα ε, παρουσιάσω τροπολογίες σε αυτή την έκθεση, παρόλο που συμφωνώ με το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης, είναι για τη χρήση της ε, ε, τεχνολογίας πληροφορικής η τεχνολογία πληροφορικής είναι πιο, το πιο προηγμένο εργαλείο επικοινωνίας που μας συνδέει με τους πολίτες και με τα άλλα όργανα εδώ. Θα ήθελα να υπογραμμίσω λοιπόν ότι είναι η πιο στρατηγική υποδομή που έχουμε τώρα και που θα έχουμε και στο μέλλον. Άρα λοιπόν θέλω να καταστήσω σαφές ότι πιστεύω ότι μακροχρόνια δεν μπορούμε να συνεχίσουμε <clears throat> να πιστεύουμε ότι αυτή τι η πιο στρατηγική υποδομή αναθέτεται σε εξωτερικούς φορείς. Αν είναι η στρατηγική τότε πρέπει να είναι η καρδιά της δουλειά μας. Και <clears throat> αν είναι στρατηγική σημασία θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό να το έχουμε εσωτερικά, να είναι ασφαλισμένο, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό έτσι ώστε να χρησιμοποιείται ευρέως, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό έτσι ώστε οι βουλευτές που δεν είναι κατά ανάγκη χρήστες του διαδικτύου να χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο διότι είναι το μέλλον μας και θέλω εδώ να προσθέσω κάτι. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε τελικά αν αυτή η στρατηγική τύχη κατάχρησης θα πρέπει εμείς να φέρουμε την ευθύνη εσωτερικά από τον ανώτερο λειτουργό ε, πληροφόρησης της Βουλής. Νομίζω ότι ο έλεγχος όλων των ευκαιριών πώς θα, ρυθμίσει αυτό το θέμα είναι θέμα το οποίο εμεί, σαν Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών, μπορούμε να το εξετάσουμε. Σα ζητώ λοιπόν να το εξετάσουμε ει βάθο είναι θέμα στρατηγικής σημασίας, επαναλαμβάνω, και θα πρέπει από το σημείο που είμαστε να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου να γίνεται καλύτερη χρήση. Και περιλαμβάνει και την ασφάλεια, την ασφάλεια των δεδομένων, την επεξεργασία των δεδομένων, όλα αυτά πρέπει να ε, αναλυφθεί η ευθύνη εντός του Κοινοβουλίου. Δεν μπορούμε να το αναθέτουμε εκτός και βλέποντα ε, τη συζήτηση για την επεξεργασία και την προστασία των ε, δεδομένων, πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ηγείται, να δείχνει τη βέλτιστη πρακτική στο θέμα αυτό. Αυτό ήταν το θέμα που ήθελα να θίξω. Αλλιώ ε, συγχαίρω του συζητητέ, Νομίζω κάθε χρόνο κινούμαστε προ τη σωστή κατεύθυνση, αλλά εδώ <clears throat> θα πρέπει να κοιτάξουμε αυτό το θέμα, διότι είναι στρατηγική σημασία. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφος κ. Φέλνερ, έχει λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή η έκθεση. Δεν έχω πολλά να προσθέσω στα όσα υπόθηκαν. Ούτε στην έκθεση. Ο κύριος Ιταλά αναφέρθηκε στις σημαντικότερες ιδέες. Ε, δημιουργείται η εντύπωση ότι κάθε χρόνο υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα που προσελκύει την προσοχή, αν είναι ένα κτίριο στο Στρασβούργο ή κάτι άλλο είναι ένα μεγάλο παράδειγμα αδικίας ή προβληματικό που προβάλλεται. Φέτος νομίζω ότι της μόδας θα είναι η ασφάλεια. Κατά την ακρόση με τον Κλάους Βέλλερ ήταν ενδιαφέρον το πώς απάντησε στις ερωτήσεις για την επίθεση στην τράπεζα. Ήρθε να επισκέπτης από τη Ουάσιγκτον και είπε ότι στη Ουάσιγκτον βλέπει κανείς Πόσο σημαντικό είναι ένα θεσμικό όργανο όταν είναι πολύ δύσκολο να μπει. Όσο πια είναι ο θεσμό στην Ουάσιγκτον, μάλλον αντιστρόφως ανάλογη σημασία του ιδρύματο του θεσμού με την ε, ε, σημασία που έχει. Δηλαδή τελικά υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία εδώ πέρα για να καταφέρεις να σου επιτρέψουν να μπει την πρώτη φορά, αλλά μετά η ασφάλεια είναι σε χαμηλό επίπεδο. Η έκθεση καλύπτει πολύ καλά το θέμα της ε, ασφάλειας. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη πραγματική ασφάλεια. Ε, με τρόμο είδα ότι είχαμε 900 φρουρούς. Τι κάνουν οι 900 φρουροί. Και κάτι άλλο που ήθελα να θέσω. Είναι πολύ καλό το ότι ο εισηγητής ασχολείται με τις περσινές επικρίσεις για το βραβείο δημοσιογραφίας. Ε, και αυτή η τάση που έχουμε να κερδίζουμε πόντους δίνοντας βραβεία. Δίνουμε πολλά βραβεία. Δεν ξέρω αν το 2011 ε, μεγαλύτερο καθήκον του νομοθετικού οργάνου θα είναι να ε, δίνει βραβεία. Θυμάμαι κάποτε που είχαμε χρόνο, γιατί δεν ομοθετούσαμε τόσο πολύ. Τώρα έχει αλλάξει η κατάσταση. Δεν έχουμε τόσο χρόνο για τα βραβεία. Τώρα για το δικό μας κανάλι, το web και για την τηλεόραση στο διαδίκτυο, το web TV και για τις δημοσιογραφικές μας φιλοδοξίες. Πολύ συχνά ε, δημοσιογράφοι του Κοινοβουλίου τηλεφωνούν στους ευρωβουλευτές και ρωτούν ποιες είναι οι απόψεις μας. Δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό. Δηλαδή πόσος κόσμος παρακολουθεί αυτό το κανάλι τελικά στο διαδίκτυο. Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές κάρτες των μελών, αυτά που αναφέρονται είναι λογικά. Θα πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που περιέχονται. Το νόημα ύπαρξης αυτής της κάρτας είναι να μας επιτρέπει να μπαίνουμε στο κτίριο. Πρέπει να σκεφτούμε όμως τι συμβαίνει με την συλλογή στοιχείων. Αν θα συλλέγονται στοιχεία όταν μπαίνουμε βγαίνουμε από το κτίριο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και τους σκιώδης για το θέμα. Δύο παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω, αν μου επιτρέπετε, και μια ερώτηση προς τον κύριο Ίτελ. Πρώτη παρατήρηση. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εδώ στην απαλλαγή φέρουμε ιδιαίτερο ε, βάρος ευθύνης. Γιατί το θεσμικό όργανο δίνει απαλλαγή στον εαυτό του ουσιαστικά. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ συνετοί, αλλιώς ε, είμαστε εκτεθειμένοι στην υποψία ότι ευλογούμε τα γένια μας. Και αυτό που μας νοιάζει είναι να καλοπερνούμε οι και όχι οι οικονομίες. Πολύ καλά το χειρίζεται ο κύριος Ήταλα και θα ήθελα να καλέσω τους συναδέλφους εδώ να ε, ενισχύσουμε πάρα πολύ το εξής σημείο. Όλοι εκείνοι που ασχολούνται και με την πολιτική προπολογισμό γνωρίζουν ότι ε, θα είμαστε σε μεγάλη πίεση για το 2011 και για τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου. 12 διορθώνει ο μιλητής, όχι για το 11, για το 12, για το χρόνο και για το Κοινοβούλιο. Και μας παρακολουθούν όλοι πολύ στενά. Σε σχέση με αυτό λοιπόν, ε, είναι σωστό αυτό που ζητάει στην παράγραφο 99 ο κύριος Ήτελε. Να δούμε, να υπολογίσουμε πόσο μας κοστίζουν οι τρεις έδρες και το μπαλάκι αυτό να το στείλουμε στο Συμβούλιο. Γιατί κάνουμε αυτό το τσίρκο, το πλανόδιο, εν πάση περιπτώσει. 160 εκατομμύρια ευρώ κοστίζει το όλο εγχείρημα. Γιατί το Συμβούλιο δεν μας επιτρέπει να κάνουμε αυτές τις οικονομίες. Να το συζητήσουμε μαζί τους. Αυτοί κάθονται στο γιου στους λήψεου, δεν πάνε πουθενά και μα φωνάζουν να κάνουμε οικονομίε. Ορίστε οικονομίε. Με ένα σμπάρο 160 εκατομμύρια ευρώ. Πώ σα φαίνεται. Εντάξει, ωραία τα χαρτιά, οικονομία στο χαρτί, αλλά αυτό είναι ψαγόνα στον ωκεανό. Πιο γρήγορη οικονομία από αυτά τα 160 εκατομμύρια δεν θα μπορούσαμε να βρούμε. Να τα πούμε σε αυτούς τους κυρίους που κάθονται πάντα στο ίδιο κτίριο. Άλλο θέμα τώρα. Τι είναι επίκαιρο και τι δεν είναι να συζητήσουμε και τα δημοσιογραφικά βραβεία και ό,τι άλλο θέλετε και για τον οίκο της ευρωπαϊκής ιστορίας. Λίγο ηρωνικά τα βλέπω όλα αυτά στην πολιτική μου ομάδα και το αναφέρω ως Hans Gert Pöttering Memorial αυτό το ίδρυμα. Τώρα αυτή τη στιγμή τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια μας χρειάζεται αυτό. Μας χρειάζεται να γίνει εδώ. Το κτίριο Eastman το θεωρώ τελείως ακατάλληλο. Χρειάζονται και πάρα πολλά έργα ε, για να γίνει μουσείο αυτό το κτίριο. Και θα κάνω και τροπολογίες, όπως είπε και κάποιος άλλος συνάδελφος. Ερωτώ τώρα τον συνάδελφο Ήτολε. γιατί δεν το κατάλαβα πάρα πολύ καλά, τι εννοείται. Την ηλεκτρονική υπογραφή παρουσίας. Εγώ είμαι νέο μέλος αλλά με την ευρωπαϊκή πολιτική ασχολούμαι εδώ και καιρό. Έχω δουλέψει και ως βοηθός εδώ που είχαμε απουσιολόγια στις εισόδους του Κοινοβουλίου και δυστυχώς κάποιοι συνάδελφοι ερχόντουσαν με τη βαλίτσα, υπέγραφαν και χαίρεται. Παίρνανε δηλαδή έτσι την ημερήσια αποζημίωση και επιτόπου έφευγαν από το Κοινοβουλίο στη Γερμανία τέτοιοι βουλευτές παρακολουθήθηκαν, μαγνητοσκοπήθηκαν, τους έδειξε τηλεόραση και η ζημιά για το κοινοβούλιο ήταν μεγάλη. Τεράστια. Λόγω της συμπεριφοράς αυτών των συναδέλφων. Στη Γερμανία χρόνια ολόκληρα χρειαστήκαμε για να φύγουμε από αυτή την εικόνα. Υποθέτω ότι και στις άλλες χώρες κάτι αντίστοιχο θα συνέβη. Το ήξεραν οι πάντες, είχαν δει τις εικόνες στη τηλεόραση. Σήμερα ακόμα καμιά φορά μας το αναφέρουν. Και οδήγησε στο γεγονός ότι φτιάξαμε αυτό το κεντρικό μητρό που είναι στα έγκατα του Κοινοβουλίου και όχι στην είσοδο, τουλάχιστον ε, θα πρέπει να διανύσουν κάποια απόσταση και να υπογράψουν και να ξαναφύγουν, γιατί και αυτό συμβαίνει, αλλά όχι στην είσοδο. Και τώρα εσείς προτείνετε ηλεκτρονική ψηφο, ε, συγγνώμη, υπογραφή ως ένδειξη παρουσίας. Κάποιος που δεν έχει μεγάλη εξοικείωση, ε, αλλά που χρησιμοποιεί ε, την τεχνολογία αυτή. Δεν μπορεί να καταλάβει και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ε, πώς θα γίνει αυτό και με τι μηχανήματα για να είμαστε βέβαιοι ότι είναι κάποιος παρόν στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου για να υπογράψει ηλεκτρονικά. Γιατί στην περίοδο του ίντερνετ η ηλεκτρονική υπογραφή σημαίνει πολλά και μακρινά. Θα ήταν ενδιαφέρον να το συζητήσουμε αυτό. Ίσως ηλεκτρονική ε, υπογραφή να μπορεί να συνδεθεί με την ηλεκτρονική είσοδο και έξοδο. Δηλαδή να ανοίγει ο βουλευτή με την κάρτα του την πόρτα για να μπει στο κοινοβούλιο. Αλλιώ έχω μεγάλες αμφιβολίες. Σα ευχαριστώ. Ο κύριο Οντί έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αναφερθώ μόνο για την παράγραφο 99 στη συνεδρία πολιτικής μας ομάδα θα ζητήσω από τον εισηγητή να μειώσει κάπως τον τόνο της διατύπωσης. Θα ήθελα, ε, εδώ εκφράζεται το αίσθημα απελπισίας αν θέλετε και ο παράδοξος χαρακτήρας του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζονται τα πράγματα. Κατανοώ την αντίδραση, ε, κυρία συνάδελφε, αλλά σε αυτές, σε αυτές τις γραμμές, σε 7 γραμμές να γράψετε τρεις αναλήθειες να γράψετε πράγματα που είναι λάθος, νομικά σημεία ασφαλμένα, δεν μπορεί να οδηγεί άσκηση πολιτικής, δεν ασκείται έτσι η πολιτική. Πρώτη γραμμή, να διαθέτουμε μόνο έδρα. Ε, ε, έχει μόνο μία έδρα το Κοινοβούλιο. Είναι το Στρασβούργο η έδρα του Κοινοβουλίου. Πρώτο σφάλμα. Γιατί αναφέρει οικονομίας. Μετά, 160 εκατομμύρια ευρώ διασπαθίστηκαν ε, ε, αν μείνουμε στις Βρυξέλλες θα κάνουμε οικονομία σε σχέση με συνεδριά στο Στρασβούργο και το ίχνος ε, του άνθρακος θα είναι χαμηλότερο στις Βρυξέλλες από το Στρασβούργο. Το ίδιο θα είναι. Η μεταρρύθμιση της συνθήκης των συνθήκων. Αυτό αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό δεν είναι αληθινό. Η συνθήκη είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και το, Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη. 27 ναι χρειάζονται. Λοιπόν, α το εξετάσουμε το πολιτικό θέμα της έδρας. Αλλά αυτό δεν αφορά το ε, Ευρωπαϊκό Συμβουλίο. Έχει δικαίωμα πρωτοβουλία για τη μεταρρύθμιση των συνθήκων. Αλλά η συνθήκη δεν τροποποιείται από τα κράτη-μέλη. Η μεταρρύθμιση των συνθήκων δεν είναι αρμοδιότητα ευρωπαϊκή. Είναι αρμοδιότητα των ε, κρατών μελών. Προσέξτε και κάτι άλλο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίση έχει δικαίωμα πρωτοβουλία στον φάτη τη μεταρρύθμιση των συνθήκων. Δεν είναι μόνο το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο, είναι η καινοτομία τη συνθήκη τη Αβώνα που ίσω διέφυγε από τα μέλη. Α διεξαχθεί λοιπόν μια πολιτική συζήτηση για την έδρα αντί να έχουμε τέτοιου είδου τροπολογίε με τόσα λάθη. Ας ασχοληθούμε με το θέμα λοιπόν της πολιτικής της έδρας. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα στη Φραγκφούρτη, το, γραφείο των διπλωμάτων της τεχνίας ε, ε, στο Μόναχο, στο Λονδίνο, η υπηρεσία φαρμάκων, τα ταξίδια, το ίχνος του φάρμακος. Έχουμε μια εβδομάδα ε, των, ε, εκλογών, 13 αποστολές του Κοινοβουλίου. Αν θέλουμε να κάνουμε οικονομίες, ασχοληθούμε όλα αυτά τα θέματα. Σαν Γάλλος λοιπόν θέλω να πω ότι αυτού του είδους μάλλον θα ήθελα να μπούμε σε διάλογο. Για να δούμε στην Ολομέλεια λοιπόν να, αν θα υπάρξει τροπολογία αυτό το θέμα γιατί ενδιαφέρει όλη την Ολομέλεια και θα πρέπει να ετοιμάσουμε μια διατύπωση που να υποσκάπτει λιγότερο την Επιτροπή μας. Είναι ένα πραγματικό θέμα. Οι πολίτες έχουν προσδοκίες και στη Γαλλία εξάλλου και στη Γαλλία. Αλλά ε, ας προσεγγίσουμε το θέμα με έναν τρόπο λογικό, ε, πραγματιστικό ε, και όχι έτσι με αυτόν τον τρόπο με μια διατύπωση η οποία είναι κακή. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Μπρεσμπάτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το συνάδελφο. Και βλέπουμε αυτή την έκθεση όχι από πλευρά λογιστική, αλλά προσπαθεί να βρει δυνάμει εξοικονομήσει στη λειτουργία του Ευρωκοινοβουλίου. Είχα κάποια σχόλια, μερικά έχουν αναφερθεί, μόνο δύο μικρά σχόλια σχετικά με την πρόσβαση στο κτίριο. Βλέπω το θέμα τη ασφάλεια, το επίπεδο ασφάλεια. Όλοι το συζητάμε εδώ και αρκετό καιρό. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να το βελτιώσουμε. Το δεύτερο επίπεδο και θέμα είναι η οικονομική προσέγγιση. Σω θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε και τις ημερήσιες συνεισφορές στην ασφάλεια. Σίγουρα οι ευρωβουλευτές μας θα πρέπει να χρησιμοποιούν ηλεκτρονική ταυτότητα για πρόσβαση στα κτίρια και υπάρχει και θέμα πιθανής πυρκαγιάς, διότι η ασφάλεια θα πρέπει να γνωρίζει πόσα άτομα βρίσκονται στο κτίριο. Είναι ε, στάνταρτ απαιτήσει αυτές. Και αυτό το σύστημα δουλεύει στη Τσεχία όχι μόνο στο κτίριο του Κοινοβουλίου, αλλά και σε άλλα κτίρια ε, και δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα. Δεύτερο θέμα. έχουμε, είναι πληροφορίες για τις, την παρουσία των βουλευτών μέσα στο κτίριο και βέβαια ε, μπορούμε να το συζητήσουμε. Χρησιμοποιούμε ε, αυτό για τα πρακτικά, διότι έχουμε κατάλογο παρουσιών για τις ε, συνεδριάσεις, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Κάτι άλλο το οποίο έχει εισηγηθεί είναι η εγώ δούλευα στον τομέα της πληροφορικής, προτού γίνω μέλος του Ευρωκοινοβουλίου, έλεξα όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται στους ε, ευρωβουλευτές. Είναι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, αλλά δεν ε, μπορούμε να είμαστε σε όλες τις συνεδριάσεις με τα notebooks, διότι δεν μας το επιτρέπουν οι δυνατότητες ε, διασύνδεσης. Θα πρέπει να ενισχύσουμε βέβαια τους εξοπλισμούς πληροφορικής, να έχουμε καλύτερα συστήματα Wi-Fi και στα γραφεία μας, εάν τότε είναι αυτός ο τόπος που πρέπει να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ιταλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους για τα σχόλια σας. Πολλά είναι σχόλια με τα οποία συμφωνώ. Αυτά που άκουσα για τα ποδήλατα, για ε, το χαρτί και τη χρήση χαρτιού. Θα σημειώσω αυτά τα σχόλια. Μιλήσαμε για την οικονομική κρίση και την εισαγωγή αυτού του σημείου στο κείμενο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, πρέπει να δηλωθεί αυτό ρητός και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσει τι μπορεί να γίνει στο θέμα αυτό. Γιατί σε κάθε κράτος μέλος οι πολίτες μας υποφέρουν, υφίστανται πιέσεις Γι' αυτό το λόγο πρέπει και εμείς να δούμε πώς δαπανώνται τα χρήματα στα θέματα πληροφορικής, τεχνολογίας των ε, πληροφοριών. Δεν είμαστε ε, και ε, πολύ αυτού του τομέα, αλλά και εγώ θα ήθελα να έχουμε καλύτερη στήριξη πληροφορικής. Έχουμε ένα νέο δίκτυο που ξεκινάει, το χρειαζόμαστε. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία κρεμούν όμω. και υπάρχει πολύ περιθώριο βελτίωσης. Αν πάμε τη χρηματοδότηση για θέματα πληροφορικής, θα ταπανώνται μεγάλα ποσά στον τομέα αυτό. Αλλά ένα μεγάλο μέρος είναι, αναθέτεται σε εξωτερικούς φορείς και νομίζω δαπανούμε πολλά στις αναθέσεις, ε, στις εξωτερικές αναθέσεις. Θα μπορούσαμε να αναθέσουμε και εσωτερικά ένα μεγάλο μέρος. Συμφωνώ με τις εισηγήσει για τροπολογίες στο θέμα αυτό και χρειαζόμαστε βελτίωση Για την ηλεκτρονική υπογραφή θέλω να είμαι πιο σαφής εδώ στο θέμα αυτό. Αυτό που θα ήθελα είναι κάθε φορά που οι βουλευτές μπαίνουν στο κτίριο να υπογράφουν με την κογκάρδα τους, με την, καρτέλα, με την κάρτα, την ε, ηλεκτρονική. Να μην περνάνε απλά από ένα διάδρομο. Οποιοςδήποτε μπορεί να περάσει από εκεί. Οποιοςδήποτε μπορεί να περάσει κατευθείαν μέσα στο χτίριο. Αλλά γιατί να μην είμαστε σαν τους άλλους. Γιατί να μην ε, βάζουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα στο σύστημα έτσι ώστε να ανοίγει η πόρτα και να καταγράφεται η παρουσία μας στο κτίριο έτσι ώστε αν προκύψει κάποια πυρκαλιά να γνωρίζουν ποιοι είναι μέσα στο κτίριο. Αυτές οι πληροφορίες δεν θα δοθούν στον τύπο, δεν θα γίνει γνωστό ποιο βουλευτής μπαίνει και ποιο φεύγει. Νομίζω Πολλοί φοβούνται αυτού του είδους διαρροές στον τύπο. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός και δεν θα συμβεί αυτό. Εάν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, νομίζω θα έχουμε πιο αποτελεσματική ασφάλεια. Ίσως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε τις ε, κάρτες ψηφοφορίας όταν μπαίνουμε στις αίθουσε, να τις βάζουμε στις μηχανές και να υπογράφουμε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί όταν υπογράφεις σε χαρτί θα πρέπει να πας πίσω και να, να, πας, ε, ε, να δεις ότι υπάρχει ένα γραφείο όπου ο κόσμος δουλεύει με απειρχιωμένο τρόπο. Θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη χρήση των πόρων, να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους μας πιο ευφυώς με την ηλεκτρονική υπογραφή. Δεν είναι δυνατό να γίνεται παντού. Βέβαια, αν πας σε κάποια αποστολή θα πρέπει να υπογράψεις το χαρτί. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα πλήρως ηλεκτρονικό σύστημα. Αυτή ήταν η ιδέα μου όμως. Ε, το Κογκρέσο στη ΣΥΠΑ το εφαρμόζουν και σε κρατή-μέλη εφαρμόζεται αυτό το σύστημα. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην μπορούμε εμείς να το εφαρμόσουμε εδώ. Τώρα, στο θέμα των τριών εδρών. Διαφωνώ με τη δήλωση ότι είναι νομικό ε, λανθασμένο. Έχουμε τρεις έδρες, όντως έχουμε τρεις έδρες και λειτουργούμε στο Στρασβούργο, λειτουργούμε στο Λουξεμβούργο και εδώ στις Βρυξέλλες. Δεν βλέπω ποιο είναι το νομικό λάθος. Τώρα για το ποιος παίρνει ε, την απόφαση λέει ότι είναι το Συμβούλιο, αλλά σε παρένθεση λέει τα κράτη-μέλη. Και σχετικά με το κόστος, είναι διοικητικό το κόστος. Τώρα, αν υπάρχει κάποιο νομικό σφάλμα εδώ, ε, θα ήθελα να το ελέγξουμε την νομική υπηρεσία και να το διορθώσουμε και να ε, κάνουμε ένα διάλογο εδώ. Αλλά ε, προσπαθούμε να ρίξουμε το μπαλάκι στο Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα πρέπει να έχουμε μια συζήτηση στο θέμα αυτό. Το Συμβούλιο ζητάει το Κοινοβούλιο να εξοικονομήσει χρήματα και εμείς μπορούμε να πούμε στο Συμβούλιο «Κοιτάξτε, αν εσεί τα κράτη-μέλη αποφασίσετε, εμεί μπορούμε να κάνουμε την εξοικονόμηση. Αλλά είμαι ανοιχτό για συζήτηση του θέματο και σίγουρα δεν ε, επιθυμώ αυτό το πράγμα να ε, μην είναι νομικό ορθό. Αλλά θα διαφωνούσα γιατί νομίζω δεν υπάρχει κάποιο νομικό σφάλμα εδώ ούτε ε, ως θέμα αρχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ιταλά. Πάμε λοιπόν στο άλλο σημείο της ημερήσιας διάταξης που αφορά την απαλλαγή 2009 στο Συμβούλιο και στα λαθεσμικά όργανα. Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή, να σας πω ότι εδώ και μερικές μέρες συναντήθηκα με εκπροσώπους τη Ουγγρική Προεδρίας κατόπιν αιτήματό τους και συνάντησα τον Υπουργό, τον Αρμόδιο τον που ήθελε να μου αναφέρει το πόσο πρόθυμη είναι η Ουγγρική Προεδρία να καταλήξει σε διοργανική συμφωνία με το Κοινοβούλιο και να σημειωθούν σημαντικά βήματα πρόοδου σε σχέση με την αποτελμάτωση που έχουμε τώρα όσον αφορά την απαλλαγή και τις πληροφορίες που χρειάζεται το Κοινοβούλιο για να διαθέσει την απαλλαγή. Εγώ δέχτηκα θετικά αυτή την κίνηση της συνεργασίας και της προσπάθειας επιτάχυνσης της διαδικασίας που παρουσίασε ο Υπουργός και δημιούργησε ήδη μια ομάδα εργασίας η Ουγγρική Προεδρία και έχει προτίθεται να έρθει εδώ στις 28 Φεβρουαρίου ο Υπουργός στην Επιτροπή μας και να αναφερθεί στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίτευξη διοργανικής συμφωνίας. Εγώ άκουσα και υπογράμμισα, επανάλαβα τη θέση μας, τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την διαδικασία της απαλλαγής. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν καλό να περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις των προσπαθειών της Ουγγρικής Προσπαθίας Προσπάθησα να παρακολουθήσουμε όλοι μας με μεγάλη προσοχή. Θα δώσω το λόγο τώρα στον συνάδελφο Ριβελίνη που είναι συγγητής αυτού του σημείου της διάταξη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η απαλλαγή των άλλων θεσμικών οργάνων συμπεριλαμβάνουν 7 ε, ειδικέ προτάσεις που αφορούν 7 ξεχωριστά θεσμικά όργανα. Αν επιτρέπετε, εγώ δεν θα ήθελα να ακολουθήσω χρονολογική σειρά, διότι ανάμεσα στα 7 αυτά όργανα υπάρχουν κάποιοι πιο σημαντικοί φορεί και είναι η έκθεση για την απαλλαγή στο Συμβούλιο, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος πριν, και υπάρχουν άλλες απαλλαγέ που έχουν μικρότερη δυσκολία. Λοιπόν, αν ο Πρόεδρος ε, μου επιτρέπει, θα ήθελα να ακολουθήσω μια διαφορετική χρονολογική σειρά. Θα ξεκινούσα από τον Γενικό Προϋπολογισμό για την προστασία, τον Φορέα Προστασίας Δεδομένων, των Ευρωπαϊκών είναι ίσονο σημασία αυτός ο φορέος που δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, η κρίση είναι θετική, είναι ικανοποιητική κατάσταση, αν και υπάρχουν κάποια προβλήματα, κυρίως το σημείο 8 της εκθέσεώς μου, αναφέρομαι στην ανάγκη να εντοπιστούν σύντομα και άλλες διοικητικά μέτρα που θα επιτρέψουν στα ε, θεσμικά όργανα να συμμορφωθούν με τις συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου. Πιο συγκεκριμένα την ανάγκη να υπάρχουν συστήματα εκ των υστέρων επαλήθευσης, ξεκαθαρίζοντας επίσης την ανάγκη να αναφέρεται πότε τέτοια αρμοδιότητα θα πρέπει να ανατεθεί. Πέρα από αυτού, στην πρότασή μου, στο σημείο 13, ε, ανέφερα ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Προστασία των Δεδομένων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην επόμενη έκθεση ετήσια δραστηριοτήτων για τη χρήση 2010 ένα κεφάλαιο που θα παρέχει απολογισμό της συνέχειας που δόθηκε κατά τη διάρκεια του έτους στις αποφάσεις της απαλλαγής ε, που έδωσε το Κοινοβούλιο. Αλλά ε, αυτό, ε, τελικά η άποψή μας είναι θετική όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, όσον αφορά την απαλλαγή. Όσον αφορά τον Ευρωπαίο Διαμοσολαβητή και αυτή την απαλλαγή, και εδώ προέκειται περί θεσμού μικρότερη σημασία που δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα. και εδώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι θετική η τοποθέτησή μας. Όμως θα πρέπει να τονίσουμε ότι παραμένει μια δυσκολία όσον αφορά τις διαδικασίες ε, προσλήψεως των προσωρινών υπαλλήλων με συμβάσει στις ορισμένες διαρκές εάν μένει αυτό θετικό πρέπει να σημειώσουμε ότι ε, δόθηκαν πρόσφατα οδηγίες για να μειωθεί το πρόβλημα που έχει σημειωθεί. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να ενημερωθεί όσον αφορά την εξέλιξη της κατάστασης, όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάμε στην απαλλαγή της Επιτροπής των Περιφερειών. Εδώ δεν υπάρχουν ούτε ιδιαίτερα προβλήματα, ούτε ε, ιδιαίτερα σε μία προσυπογράμμιση και νομίζω ότι αυτή η απαλλαγή μπορεί να δοθεί τάχιστα. Μετά έχουμε την απαλλαγή όσον αφορά την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και αυτό ε, αυτός είναι ένα, αυτό είναι θεσμικό όργανο που δεν ε, δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες όσον αφορά την απαλλαγή και εδώ συνολική η εντύπωση είναι ικανοποιητική όμως ε, πρέπει να πούμε ότι οι απαντήσεις που η Επιτροπή έδωσε στις παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των μελών ε, κατά την ε, ταπεινή μου άποψη δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικές σε διαφοροποιώντας εδώ την κατάσταση που αφορά την Επιτροπή των ε, Περιφερειών που δεν έχει ακόμα τις δηλώσεις αλλά έκανε μια μελέτη όσον αφορά τις διάφορες επτομέρειες της προσέγγισης η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή δεν υιοθέτησε ακόμα τα σχετικά μέτρα ούτως ώστε να επιληθεί το θέμα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Τώρα κάτι άλλο που έχω να υπογραμμίσω όσον αφορά συγκεκριμένη απαλλαγή ε, είναι το θέμα που αφορά την έκθεση του κυρίου Βερμέιο Γκάρντε, πρώην υπαλλήλου της Επιτροπής, ο οποίος ε, έχει υποθεί στην Όλαφ. Ζητήθηκε κατόπιν αιτήματός μου, ζήτησα από τη γραμματεία να μας πληροφορήσει η Όλαφ στις 18 Ιανουαρίου και έλαβα απάντηση όπου η απάντηση σημείωνε ότι η υπόθεση συγκεκριμένη ακόμα περνά από μια προκαταρκτική φάση μέχρι σήμερα δεν κατέφθασε καμία ανακοίνωση σχετικά με αυτή την υπόθεση. Πιστεύω λοιπόν ότι θα ήταν καλό να αναφέρουμε στην έκθεση αυτό το γεγονός. Πάμε μετά στην απαλλαγή όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εδώ έχουμε διάφορα σημεία, μπορούμε να υπογραμμίσουμε. Πιστεύω ότι η συνολική εικόνα όσον αφορά τις επιτευχθήσεις όσον αφορά της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και τη λειτουργία ε, του δικαστηρίου γενικά γενική, η τελική συνολική εικόνα είναι θετική όμως θα πρέπει να εισημάνω κάποια πράγματα και πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβει υπόψη όλα αυτά η Επιτροπή ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις παρενέσεις του ελεκτικού συνεδρίου, ούτε να προετοιμάσει καλύτερα και να συντονίσει καλύτερα τις διαδικασίες για δημόσιες προμήθειες. Πέραν αυτού, το Κοινοβούλιο πιστεύω ότι ενδιαφέρεται αρκετά για αυτό το θέμα, δηλαδή να μειωθεί να, η αύξηση της διάρκειας των υποθέσεων και η μείωση της εξετάσεως των υποθέσεων που παρατήθηκε το τελευταίο χρόνο, αυτό είναι μια κατάσταση που πρέπει να βελτιωθεί. Ε, όμως τελικά η απόφαση όσον αφορά την απαλλαγή, η τοποθέτηση είναι θετική. Όσον αφορά το ελεκτικό συνέδριο, απαλλαγή του ελεκτικού συνεδρίου, εδώ έχουμε διάφορες παρατηρήσεις. Σαν αρχή της απαλλαγής και λαμβάνοντας υπόψη την, τα καθήκοντα του ελεκτικού συνεδρίου στα πλαίσια των θεσμικών οργάνων της Ευρώπης, εδώ πιστεύω το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό όσον αφορά ε, τις ιδιαιτερότητες και τον τρόπο λειτουργίας του ελεκτικού συνεδρίου, την αμική του ελεκτικού συνεδρίου. Οι προσπάθειες που καταβάλει τα τελευταία χρόνια το ελεκτικό συνέδριο για την βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων και πιο συγκεκριμένα με την εξέταση συμπληρωματικών δειγμάτων, προσθέτων δειγμάτων, είναι σίγουρα ένα θετικό γεγονός και καλούμε όμως να επεκτείνει αυτή την, ε, αυτή την πρακτική του ελεκτικού συνεδρίου να μας καλεί το ελεκτικό συνέδριο να εφαρμόσουμε και εμείς παρόμοιες τακτικές. Έχω κάτι συγκεκριμένο ε, να πω που το αναφέρω ε, στο σημείο 14 της εκθέσεώς μου. Στο σημείο λοιπόν 14 της ε, εκθέσεώς μου για την απαλλαγή αναφέρω και σε σχέση με αυτά που είδαμε στον τύπο πρόσφατα ότι υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες όσον αφορά το ελεκτικό συνέδριο ότι μπορεί να επηρεαστεί το ελεκτικό συνέδριο. Όσον αφορά αυτό το σημείο θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά σαφείς. Θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο όπως και στο άρθρο 14 αναφέρω της απαλλαγής μου, να υπογραμμίσουμε ότι το ελεκτικό συνέδριο ε, ε, δεν επηρεάζεται και θα πρέπει να πούμε ότι το ελεκτικό συνέδριο είναι, ε, πρέπει να εξάρτητο. Και θα πρέπει να γίνει μια εμβάθυνση στον αφορά το θέμα. Υπογραμμίζουμε, λέγω, το πώς επηρεάζεται το ελεκτικό συνέδριο, η δυνατότητα που υπάρχει να επηρεάζεται και μπορούμε ίσως να δεχτούμε και κάποιες συστάσεις που ακούγονται ούτω ώστε αυτό το άρθρο 14 να τροποποιηθεί κάπως και να μην υπογραμμίζεται το ζήτημα που γεννήθηκε προ καιρού. Χρειάζεται περαιτέρω εμβάθυνση και συζήτηση από αυτού του θέματος πιστεύω διότι είναι ιδιαίτερα προβληματικό το θέμα ε, και έχει χαρακτήρα πολιτικό θα μπορούσε να πει κανείς. Τέλος, φτάνουμε στο σημαντικότερο σημείο, την απαλλαγή του Συμβουλίου που σίγουρα αντιπροσωπεύει και το πιο προβληματικό χαρτοφυλάκιο. Ε, είναι άχρηστο να σταθώ στο πόσο σημαντικό είναι οι πληροφορίες που ζητούνται να είναι διαθέσιμες ε, πλήρως και συνοπτικά και σε, λεπτομέρεια να δείτε πληροφορίες και συνοπτικά. Θα ήθελα να υπογραμμίσω όμως ε, ποια είναι η ενδεχόμενη διέξοδος όσον αφορά το μπλοκάρισμα το θεσμικό ε, το οποίο αντιμετωπίζουμε εδώ και αρκετά χρόνια. Το υπογράμμισε πριν ο Πρόεδρος ότι καταβάλλεται μια προσπάθεια της ε, Ουγγρικής Προεδρίας και ο ο Ούγκρος ήρθε να με επισκεφθεί για να με ενημερώσει για τα βήματα τα οποία κάνουν οι Ούγγροι για να αποφευθεί το μπλοκάρισμα και πιστεύω ότι από αυτή την έποψη η δουλειά που κάνουμε για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια δίνει ένα ρόλο εντελώς διαφορετικό στο Κοινοβούλιο και όλα αυτά που συμβαίνουν πιστεύω ότι είναι πολύ θετικά αν συμφωνεί ε, και ο Πρόεδρος για το ρόλο που καλείται να διαταματήσει το Κοινοβούλιο σε αυτή τη φάση. Το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε, κυρίως όσον αφορά το σημείο 8 της απαλλαγής μου και την έκθεση που ετοιμάσαμε τους κοιόδης ηγητές την περασμένη εβδομάδα. Είναι δυνατόν να βρεθεί μια διέξοδος όσον αφορά, να μπορέ... όσον αφορά την απαλλαγή για να μπορέσουμε να χορηγήσουμε την απαλλαγή και ή δυνατόν επιπίας βάσεως πρέπει να κινηθούμε για τις ε, διαπραγματεύσεις. Εγώ πιστεύω ότι τα σημαντικά σημεία είναι τα ακόλουθα. Ε, βέβαια, διάκριση μεταξύ διαδικασίας προπολογισμού και διαδικασίας απαλλαγής. Η πρόσβαση στα έγγραφα από πλευράς του Κοινοβουλίου, τα οποία είναι σημαντικά για το σκοπό της απαλλαγής. Επίσημες επαφές μεταξύ της Επιτροπής μας και της Γενικής Γραμματείας και της Προεδρίας ούτως ώστε να διεξάγονται οι συνομιλίες στο Κοινοβούλιο. Απαντήσεις γραπτές από το Γενικό Γραμματέα στις ερωτήσεις που διατυπώνει το Κοινοβούλιο. Εάν όλα αυτά τα συμμερίζεται η Επιτροπή μας, θα πρέπει να θέσουμε και ένα μεταγενέστερο ερώτημα τι είμαστε διατεθειμένοι να παραχωρήσουμε για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα αίσιο τέλος όσον αφορά στις διαπραγματεύσεις. Παραδείγματο χάρη, το αίτημα πρόσβαση στα έγγραφα του Κοινοβουλίου που κατά την ταπεινή μου άποψη είναι εσφαλμένο από πλευράς του Συμβουλίου διότι δεν μπορεί να είναι κάτι ανεφόρον και λόγω του πολιτικού ρόλου και της διαφορετικής σημασίας που έχουν τα διοθεσμικά όργανα. Είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Πώς το βλέπουμε. Και το αίτημα του Συμβουλίου τ' άλλο. Το αίτημα μάλλον αυτό δεν είναι σε αντίθεση με το άρθρο 319 των συνθήκων που αναγνωρίζει πράγματι στο Συμβούλιο το δικαίωμα να μπορεί να κάνει συστάσεις αλλά θέτει τα δύο θεσμικά όργανα επί διαφορετικών βάσεων, σε διαφορετική θέση. Άρα ήδη το άρθρο 319 της συνθήκης που είναι το άρθρο που κατά κάποιο τρόπο το Συμβούλιο προβάλλει στις συζητήσεις είναι ένα όπλο υπέρ του ε, Συμβουλίου αλλά αποτελεί και μια διευκρίνηση ε, όσον αφορά τι, απάντηση πρέπει να δώσουμε στο Συμβούλιο. Είναι σημαντικό σημείο. Ασχολούμαστε με ένα θέμα επιτέλους που επί σειρά ετών ανεβάλλεται και δεν επελίετο. Το θέμα λοιπόν χρειάζεται βαθύ προβληματισμό από πλευράς όλων μας. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει ανάγκη μια άλλης συνάντησης με τους σκιώδεις εισηγητές. Υπάρχει ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης σε συζητήσεις με τον Πρόεδρο, διότι σε αυτή την απαλλαγή παίζουμε ένα ρόλο που έχει μεγάλη πολιτική σημασία. Αυτή η απαλλαγή έχει μεγάλη πολιτική σημασία όσον αφορά τη λειτουργία, τα καθήκοντα, τη σημασία που έχουν τα διάφορα θεσμικά όργανα, τον κεντρικό ρόλο του Κοινοβουλίου που αποτελείται από δημοκρατικά λεγμένα μέλη, από μια αρχή που είναι διαφορετική και μεγαλύτερη από τα άλλα θεσμικά όργανα. Έθεσα αυτά τα σημεία προς προβληματισμόν σας, παρουσίασα τις δικές μου προτάσεις όσον αφορά τις επτά απαλλαγές και πιστεύω ότι στο τέλος αυτό το θέμα, το σημείο αυτό, που αφορά το άρθρο που αναφέρεται στο άρθρο 14 για την απαλλαγή ε, του ελεκτικού συνεδρίου είναι ε, σημείο που θα μα βοηθήσει στι περαιτέρω συζητήσει για να λύσουμε τα κρεμή θέματα. Ευχαριστώ, Λε Πρόεδρο. Ξεκινάμε λοιπόν τη συζήτηση. Συνάδελφο Αγιάλα έχει το λόγο. Ναι. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστούμε τον κύριο Ριβελίνη για την έκθεσή του και για την διαθεσμότητά του να συναντηθεί με τους σκιώδες εισηγητές για να εξασφαλιστεί μια κοινή κατανόηση της θέσης του Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό. Θα ακολουθήσω τη σειρά που ακολούθησε ο κύριος Βελίνη. Φυσικά υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά για τον ε, επόπτη προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων, το διαμεσολαβητή, την Επιτροπή των Περιφερειών, αλλά ευτυχώ αυτά τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Αλλά θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου σε τρία από τα όργανα στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Ριβελίνη, τα οποία μπορεί να είναι προβληματικά. Πρώτα απ' όλα την ΕΟΚΕ, όπως είπε ο κύριος Ριβελίνη, πέραν από τα προβλήματα που σχετίζονται με τις δαπάνες ταξιδίου των μελών, υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Υπάρχει μια καταγγελία ενός από τα μέλη από τον Όλαφ το 2010 σχετικά με ε, την, μια κατάσταση της νομικής υπηρεσίας και υπήρχαν κάποιες παρατυπίες που έγιναν από τον Γενικό Γραμματέα ε, της ΕΟΚΕ. Και πάλι η Όλαφ ε, απέδειξε ότι είχε πάρα πολύ χρόνο από το Σεπτέμβριο. Στην αρχή μας είπε ότι δεν έγινε τίποτα, μετά ε, τον πήραν τηλέφωνο αυτόν που είχε κάνει την καταγγελία, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο και τώρα το ψάχνουν λένε. Εγώ θα παρακαλούσω τον κύριο Ριβελίν και την Επιτροπή μας ακριβώς επειδή υπήρξε αυτή η ολιγορία από πλευράς Όλαφ από τον Απρίλιο του 2010 και από το Δεκέμβριο τελευταία καταγγελία δεν έχει γίνει τίποτα. Λοιπόν, ε, μας λένε ότι η απόφαση δεν θα ληφθεί καταρχήν μέχρι τον Απρίλιο. Γιατί έχουμε χρόνο, λέει όλα. Ε, σας είπα ότι έγινε μια καταγγελία από ένα σύμβουλο που είναι πάρα πολύ ανισχυτική και θα πρέπει να διατηρηθεί ανοιχτό το θέμα μέχρι να μας απαντήσει η Όλαφ αν ε, ευσταθούν αυτά ή όχι. Για το ελεγκτικό συνέδριο, πολύ ωραία τα εξήγησε ο κύριος Ριβελίνη. Επιπλέον, στην Επιτροπή μας ανέκαθεν λέμε ότι θα πρέπει να βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα, μετά ρύθμιση ε, από την περασμένη θητεία τα ίδια λέμε. Τα κατάλαβε το Ελεκτικό συνέδριο, μας το έχει πει επανειλημμένος και τώρα έχουμε μια σειρά δράσεων που έχουν ε, υλοποιηθεί ή υλοποιούνται για να βελτιωθεί η λειτουργία και αποτελεσματικότητα του ελεκτικού συνεδρίου. Ε, χαίρομαι που ο κύριος Ριβελίνη ε, δηλώνει προθυμία να το κοιτάξει. Παρακαλώ και εγώ στο σημείο 14 λέω το εξής. Το γεγονός ότι υπάρχει μέλος του ελεκτικού συνεδρίου που χρόνια ολόκληρα αργότερα, χωρίς να έχει πει τίποτα προηγουμένως, μόλις φύγει, ε, παραβιάζει και το επαγγελματικό απόρριτο που πρέπει να το χαρακτηρίζει και που οφείλει να τηρεί και μπαίνει σε κατηγορίες αφήστε δε που είναι και προσωπικές αυτές αντιπαλότητες. Να μην διωγγώσουμε εμείς το πρόβλημα, να το διαλευκάνουμε. Στο σημείο 14 λοιπόν, να κοιτάξουμε αυτό που μας ενδιαφέρει, να κάνει καλύτερα τη δουλειά του, δηλαδή το ελεκτικό συνέδριο, όσο γίνεται μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, να δουλεύει καλά και να αυξάνει την αποτελεσματικότητά του και αν χρειαστούν και μεταρρυθμίσει. Και εμεί συμφωνούμε και συνεργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό θα προτιμούσα. Και να μην δίνουμε την εντύπωση ότι κάποιοι προχωρούν σε ξεκαθάρισμα λογαριασμό, ότι ξαφνικά ξύπνησε το κοινοβούλιο και ανακάλυψε προβλήματα. Μα το διάλογο που έχουμε εδώ και χρόνια το απαιτούμε και υπάρχουν και βελτιώσεις. Μπορεί να μην είναι αρκετέ, αν δεν είναι να αυξηθούν. Για το Συμβούλιο τέλος συμφωνώ με αυτά που λέει ο κύριος Ριβελίνη για τη στρατηγική σημασία του ρόλου του Κοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά τη διοργανική ε, σχέση και συμφωνία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, Κοινοβουλίου, ε, έχει μεγαλύτερη σημασία πια αυτό το θέμα. Και θα παρακαλούσα το εξή. Αντί να διερωτώμαστε... Μακρηγορώ, ε. ε, ε, ε λοιπόν, αντί να α, τι παραχωρήσεις είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε προς την κατεύθυνση αυτή, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι αν μέχρι σήμερα το Συμβούλιο, όχι η Ουγγρική Προεδρία, που δεν την αμφισβητώ καθόλου την καλή της πρόθεση και θα χαρούν πολύ και τα λοιπά και εμείς θα χαρούμε να συνεργαστούμε και ό,τι άλλο θέλετε και να αποκατασταθεί η ε, νομιμότητα, η θεσμική νομιμότητα και ομαλότητα στη σχέση μας με το Συμβούλιο. Είναι το μόνο που δεν έχει απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Και από πέρσι το έχει αναγνωρίσει η Ισπανική Προεδρία στα διοργανικά και στη διακυβερνητική συνεργασία. Βιασύνη δεν υπάρχει, μεν. Το Κοινοβούλιο θέλει περισσότερα και ανεξάρτητα από την ε, καλή πρόθεση της Ογκρικής Προεδρίας, την οποία καθόλου δεν αμφισβητώ, θα πρέπει να λυθούν αυτά τα θέματα. Και δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε θέματα ήδη παραχωρήσεων ή υποχωρήσεων. Όχι, να δούμε τι έχει κάνει το Συμβούλιο μέχρι τώρα. Τι απαντήσεις μας έχει δώσει γραπτός στο ερωτηματολόγιο. Και τι πετύχαμε συγκεκριμένα. Νομίζω δεν είμαστε σε θέση τώρα να εκφράζουμε ικανοποίηση, ούτε να μιλάμε για υποχωρήσει και παραχωρήσει. Να μπούμε στην ουσία των θεμάτων με μεγαλύτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα που θα πρέπει πάντα να απαιτεί το Κοινοβούλιο και όχι να κάνουμε βήματα πίσω. Ανεξάρτητα από τα στοιχεία του προπολογισμού που έχει άλλες αρμοδιότητες πλέον το Συμβούλιο. Αλλά το άρθρο 319 τους ε, αναγνωρίζει δικαίωμα συστάσεων. Ξέρουμε τι είναι συστάσεις. Δεν είναι επιβολές, ε, ε, επιταγές, δεν είναι διαταγές, δεν είναι τίποτα, είναι συστάσεις. Όχι λοιπόν πιστοδρόμηση, κύριε Λιβερή, είναι πολύ νωρί να μιλάμε για υποχωρήσεις και παραχωρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ να επενθυμίσω τους συναδέλφους ως πολιτικοί συντονιστές σε αυτή την Επιτροπή αποφασίσαμε να καλέσουμε σε ξεχωριστή συνεδρίαση και τον Πρόεδρο Καντέρα του Ελεκτικού Συνεδρίου και Βεγγίρ του, ε, ε, τις επόμενες μέρες ώστε να έχουν πιο σαφές ε, πλαίσιο όσον αφορά το θέμα αυτό που είναι σοβαρό. Ο κύριος Μούλτερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ε, κάθε φορά έχουμε αυτό το θέμα της σχέσης με το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Είναι δύο σημαντικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω δεν μπορούμε κάθε χρόνο να έχουμε καυγάδες για αυτό το θέμα. Ό,τι με αφορά, το Συνοβούλιο θα πρέπει να είναι πλήρως ανοιχτό ε, για τις μεθόδους του που προς το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση να σχολιάζει ε, σχετικά με την διαχείριση του Κοινοβουλίου ε, και η αρχή που είναι υπεύθυνη για την απαλλαγή είναι το Κοινοβούλιο εμείς ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να είμαστε πλήρως ανοιχτοί προς το Συμβούλιο, μπορούν να μας επικρίνουν όσο είναι δυνατόν, αλλά το αντίστροφο επίσης θα πρέπει να ισχύει. Τώρα που έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας με την ύπατο εκπρόσωπο, ένα περίεργο μείγμα αξιωματούχου του Συμβουλίου και της Κομισιόν είναι αδιανόητο το Κοινοβούλιο να μην μπορεί να ελέγχει τις δαπάνε του Συμβουλίου στο τομέα και ΚΕΠΑ. Νομίζω είναι εντροπή που πρέπει να επαναλαμβάνουμε σε αυτό το ψήφισμα ότι ε, αυτό το πράγμα ξανά και ξανά. Πριν από χρόνια είχαμε στην ε, διοργανική συμφωνία ότι θα πρέπει να γίνονται συναντήσεις με το Συμβούλιο για να μας ε, ενημερώνουν για την ΚΕΠΑ. Αν το Συμβούλιο δεν το κάνει, αυτό αποτελεί παράβαση της συμφωνίας και δεν είναι αποδεκτό, είναι παράδεκτο. Ε, ως όργανο ε, είναι, έχει υποχρέωση για θέματα ασφάλειας και το Κοινοβούλιο το ελέγχει και θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια από πλευρά του Συμβουλίου αλλά και εμείς θα πρέπει να πούμε στο Συμβούλιο είστε πλήρως ελεύθεροι να μας επικρίνετε για οποιοδήποτε θέμα διαχείρισης, θα το λάβουμε υπόψη, η απόλυτη αρχή είμαστε εμείς για την απαλλαγή, αλλά θα πρέπει να υπάρχει η διαφάνεια εκατέρωθεν. Και θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Γκάιρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές ε, που ασχολήθηκαν με το θέμα. Χαίρομαι που είναι μεγάλη ομοψυχία μεταξύ των πολιτικών ομάδων στην Επιτροπή μας για αυτό το θέμα. Το διαπιστώνουμε. Θέλω να υποστηρίξω και να τονίσω αυτά που είπε η κυρία Γιάλα Σέντερ σε δύο σημεία. Στο ελεγκτικό συνέδριο εσείς, Πρόεδρε, ορθότατα είπατε ότι είχαμε συμφωνήσει με τους συντονιστές να ασχοληθούμε ξανά και με μεγαλύτερη προσοχή με αυτό το θέμα. Διότι το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο θα πρέπει να είναι υπεράνω πάσης υποψίας. Έκανε κάτι δηλώσεις στον τύπο ένα πρώην μέλος του ελεκτικού συνεδριού για πάγιες και παλιές πρακτικές ετών χρειάζονται αυτές οι δηλώσεις επεξεργασία για μας, για από για να βεβαιωθούμε τι είναι γεγονός, τι είναι παρανόηση, τι είναι ενδεχομένως ε, υπερβολή για τον αλφαβήτα λόγο. εμένει σε αυτές τις δηλώσει και τις αιτιάσει ε, που είδαν το φως τη δημοσιότητας στο πρώην μέλο, ή δεν θα έχει αποσύρει αυτά. Δεν θα πρέπει να κολλάνε τέτοιε υποψίες και να απλανώνται για το ελεκτικό συνέδριο. Και επειδή είναι παλιά ιστορία αυτή, δεν αφορούν όμως πλέον το έτος 2009 για το οποίο συζητούμε σήμερα για την απαλλαγή. Γι' αυτό θα έλεγα για το ελεγκτικό συνέδριο, να το λάβουμε υπόψη μας αυτό, ε, στους συντονιστές. Παρακαλέσαμε να έχουν τη δυνατότητα και οι δύο, και το πρώην μέλος αυτό και ο πρόεδρος του ελεγκτικού συνεδρίου και κατά πλειοψηφία πρότειναν οι συντονιστές αυτή τη συνεδρίαση να γίνει κυκλισμένο των θυρών. Ήρθε ο πρόεδρος Καρντέρα για, το, για την ημερήσια διάταξη. Τώρα έχουμε το πρόγραμμα εργασίας του ελεκτικού συνεδρίου. Είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει να είναι και κλεισμένο των θυρών. Μπορεί να τα πει και δημόσια αυτά. Τον τιμά. Ωραία. Να ρωτήσουμε τους δύο ενδιαφερομένους τι ε, τους ενδιαφέρει, τι ε, θα ήταν πρόθυμοι να συμφωνήσουν και παρά τα όσα είπα εγώ ε, αντίθετα στη συνεδρία των συντονιστών είμαι διατεθειμένος να γίνει αυτό και σε δημόσια ακρόαση. Για το Συμβούλιο, στο παρελθόν ήταν τελείως γελία η διαδικασία. Κανονιστική πρόταση ανήκουστη. Εγώ δεν πίστευα στα αυτιά μου όταν ανέλαβα εδώ ως βουλευτής και μου είπανε ότι η απαλλαγή βασίζεται λέει σε μια συμφωνία κυρίων το 1973 και άμα πάει κανείς να διαβάσει αυτή τη συμφωνία κυρίων δεν έχει λέξη για την απαλλαγή αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς ή των αδελφών Γκρίμα θέλετε και χαίρομαι πάρα πολύ την Ισπανική Προεδρία γιατί δεν λέει τίποτα αυτή η διοργανική συμφωνία παρά μόνο ότι ο ένας αφήνει στην ησυχία του τον άλλον για την απαλλαγή η Ισπανική Προεδρία ζήτησε μια πιο αξιοπρεπή διαδικασία. Τελικά δεν έχει λυθεί οριστικά αυτό το θέμα ούτε από τις συνθήκες ούτε από τα έγγραφα. Υπάρχουν διάφορα έγγραφα. Ε, η συνθήκη είπε και ο συνάδελφος Μολύνταρ για τη διοργανική συμφωνία. Κάποιες παραγράφους, κάτι τμηματικές ρυθμίσεις. Πρέπει να το λύσουμε αυτό. Επίσης όλοι γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι η Προεδρία. Ούτε η Ουγγρική, ούτε η Ισπανική, ούτε η Βελγική, ούτε καμία προεδρία εκάστοτε. Το πρόβλημά μας είναι ο Γενικός Γραμματέας και η διοίκηση του Συμβουλίου. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Διότι... Πώς να το πω... Ο συγκεκριμένος Γενικός Γραμματέας και η διοίκησή του ποντάρουν στο γεγονός ότι είναι αρρύθμιση αυτά και δεν θέλει να λογοδοτήσει εμάς. Εμείς δεν έχουμε καθόλου εικόνα για το πώς τηρούνται οι λογαριασμοί του Συμβουλίου. Οπότε δεν μπορώ να συμμετέχω ως βουλευτή στην απαλλαγή του Συμβουλίου. Με βάση ποια έγγραφα, αφού δεν έχω τίποτα να βασιστώ και να κρίνω και ευγνωμονώ το συνάδελφο Ριβελίνη που έχει κάνει προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή για να προχωρήσουμε. Πρέπει να ζητήσουμε ένα δρόμο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι αυτή η κατάσταση. Χρόνια ολόκληρα να διαιωνίζεται αυτό το πρόβλημα με το Συμβούλιο. Και είμαι και πρόθυμος να το συζητήσω με όποιο θέλετε. Βλέπω ευνοϊκά και τις ε, προτάσεις του κυρίου Μίλντερ να ληφθεί περισσότερο υπόψη η αμοιβαιότητα όπου χρειαζόμαστε και διαπραγματευτική εντολή της Επιτροπής μας ή δεν ξέρω ποιανού ε, διαπραγματεύεται. Και θα παρακαλούσα και θα επιθυμούσα να το ξανασυζητήσουμε τη νομική μας υπηρεσία για να μας εξηγήσουν πού τελειώνει η εντολή της ε, δημοσιονομικής αρχής που χορηγεί την απαλλαγή, τι γίνεται με τα έγγραφα του Συμβουλίου. Όπως σας είπα, εγώ τα βλέπω όλα αυτά θετικά και ευνοϊκά για μεγαλύτερη διαφάνεια. Και να αλλάξει κάποια στιγμή η διοργανική αυτή συμφωνία που πρέπει έτσι κι να γίνει καινούργια διαπραγμάτευση. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να δώσω απαλλαγή αφού δεν έχω τα στοιχεία. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Ριβελίν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να κράσω, αν έχει την καλοσύνη, μια σκέψη. Αυτή η Επιτροπή επ' αυτής της απαλλαγής, επί των διαφόρων απαλλαγών, καταφέρνει να βρει μια συνεργασία πέρα από τις πολιτικές ομάδες. Αυτή η Επιτροπή κινείται προ όφελο των Ευρωπαίων πολιτών και του Κοινοβουλίου. Πέρα από τις διαφορές που έχουμε μεταξύ μας. Και θα ευχαριστήσω του συναδέλφους Αγιάλα, Μούλτερ και Γκάιερ, διότι εν γέννη ε, συμφωνούμε όσον αφορά αυτό το θέμα. Από την τελευταία παρέμβαση θα ξεκινούσα του συναδέλφου Γκάιερ. Ε, και όπως και στη συνεδρία των προηγούμενων ε, ημερών συντονιστήκαμε στο ίδιο μήκο κύματο και εδώ το ίδιο. Είναι ουσιαστικό η συμφωνία του 1973, η, η συμφωνία κυρίων πρέπει να επανεξεταστεί. Από το 1973 μέχρι σήμερα υπάρχει άλλος κόσμος, άλλη Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να έχουμε τέτοιου είδους συμφωνία και ενδεχομένω εάν κάνουμε συμφωνία μεταξύ κυρίων και κυριών του 2011 αυτή να ε, εξεταστεί από την αρχή και τα θεμελιώδη σημεία να είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Αυτή πρέπει να είναι η αφετηρία για την απαλλαγή. Για τη συνάδελφο Αγιάλα τώρα. Να πω το εξής. Πράγματι, η προβληματική όσον αφορά την απαλλαγή της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής αληθεύει αυτός ο προβληματισμός, αλλά δεν μπορούμε. Υπάρχει διαφορά σημασίας μεταξύ των δύο ζητημάτων. Είναι εντελώς διαφορετική σημασία. Η χορήγηση της απαλλαγής ε, αποτελεί μια βάθηση όσο συνέβησαν. Πρέπει να είναι ξεχωριστά αυτά τα θέματα. Σημαντικά αυτά που θίξατε. Αλλά πρέπει να υπάρχει και ισορροπία μεταξύ απαλλαγής και εμβάθυνσης στο θέμα. Όσον αφορά το άρθρο 14 για την απαλλαγή στο ελεγκτικό συνέδριο, εγώ προετοίμασα και δεύτερη εκδοχή του άρθρου 14, λίγο πιο soft, όπως ζήτησε η κυρία Αγιάλα, η συνάδελφος της κυρία Αγιάλα. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να συναντηθούμε στη συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών και να συζητήσουμε αυτή τη νέα διατύπωση του άρθρου 14 και να βρούμε ίσως μεταξύ μας σημείο επαφής και να συμφωνήσουμε διότι καταλαβαίνω την ανησυχία της συναδέλφου Αγιάλα, είναι θεμητή. Δεν είναι κάτι φανταστικό και ανύπαρκτο. Πιθανότατα χρειάζεται ούτως η πίν να κάνουμε πιο ήπιο το άρθρο 14 της ε, εκθέσεως μου για να δώσουμε μεγαλύτερο κύρος στο ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου. Τώρα, όσον αφορά την απαλλαγή του Συμβουλίου, συμφωνώ απόλυτα με τους τρεις συναδέλφους που μίλησαν και κανείς συνάδελφε Αγιάλα θεωρεί ότι... Ε, αφισβητεί την διαπραγμάτευση. Επιτέλους αντιμετωπίσαμε αυτό το θέμα μετά από τόσα χρόνια. Και εγώ πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί λύση στο πρόβλημα. Κατά ποινή μου άποψη. Χρειάζεται η μέγιστη στεναρότηση από την πλευρά μας. Ε, βέβαια, στα πλαίσια σωστής επαφής και ισορροπίας μεταξύ θεσμικών οργάνων και στα πλαίσια βούλησης να καταλήξουμε σε έναν κοινό στόχο. Κανείς δεν ζητά να κάνουμε ένα βήμα ούτε μίνι βήμα προς τα πίσω. Αλλά όταν ξεκινά γύρος διαπραγματεύσεων και με θεσμική ευγένεια που παρουσιάζει η Ουγγρική Προεδρία η οποία ζήτησε συνάντηση με τον πρόεδρο Ντεμαζίστης που ήθελε να συναντηθεί μαζί μου η Προεδρία για να εκφράσει τη βούληση επίτευξης συμφωνίας. Με όλα αυτά πιστεύω ότι γίνεται υποχρεωτικό από την πλευρά μας να καθίσουμε σε ένα τραπέζι συζητήσεων, συζητήσεων όχι διαπραγματεύσεων, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι υπερεσπαζόμαστε τα δίκαια δικαιώματα του Κοινοβουλίου και των λαών. Αλλά θα πρέπει όταν κανείς κάθεται στο τραπέζι, σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, που ξεκινάει και που θέλει να φτάσει. Διαφορετικά, κάθεσαι σε ένα τραπέζι συζητήσεων να κάνεις τι, τι να κάνεις να φλιαρίσει. Δεν νομίζω ότι θέλουμε κάτι τέτοιο. Και έχουμε χρέο, έχει χρέο ο να παρουσιάσει τις προθέσεις του. Επαναλαμβάνω, θα πρέπει να υπερασπιστούμε στεναρά τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου, αλλά θα πρέπει να ζητήσουμε από τους συναδέλφους, από την Προεδρία να μας πούν ποιοι είναι οι όροι τη συζητήσεω. Ε, ποια παραχώρηση ενδεχομένως μπορούμε να συζητήσουμε Ποιο είναι το μέγιστο όριο των διαπραγματεύσεων της συναλλαγής. Εγώ εκπροσωπώ την Επιτροπή, αλλά θέλω να συνοψίζω, να συναθρίζω τις δικές σας θέσεις όλων. Και υποχρεούμε να θέσω σε συζήτηση αυτό το θέμα. Και μάλιστα σας ζητώ να μου δώσετε ενδείξεις, προτάσεις ε, διότι είναι σαφές πρόεδρε, το επαναλαμβάνω και το επαναλαμβάνω υπογραμμίζοντάς το ότι θέλω να είμαι μία σύνθεση, να συνοψίζω, να συναθρίζω τη βούληση της Επιτροπής και λοιπόν η Επιτροπή θα πρέπει να κατευθύνει τη δουλειά μου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Αλοκληρώσαμε, η κυρία Γιάλα κάτι να πει. Ναι, Πρόεδρε, ε, για το ελεκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ριβελίνη. Ναι, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε όλα όσα είπε. Θέλω κάτι να διευκρινίσω. Εγώ δεν θέλω πιο soft το 14, πιο μαλακή διατύπωση, αλλά ε, να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και στη σημασία των σχέσεων με το Ενακτικό Συνέδριο και του Κοινοβούλιο και είναι προσωπική περίπτωση. Ευχαριστώ, Συνέθα Γιάλα. Περνάμε σημείο 11. Ε, πρόγραμμα εργασιών 2011 του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Καλωσορίζω τον πρόεδρο Καλντέιρα ε, που μπορεί να έρθει και να πάρει τη θέση του και να πάρει και το λόγο όποτε μπορέσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής σας, κυρίες και κύριοι, είναι και πάλι τιμή για μένα, ευκαιρία που έχω να απευθυνθώ στην Επιτροπή σας, ε, κινώντας ε, τη δεύτερη θητεία μου ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Προσβλέπω πάρα πολύ να, στη συνέχιση της συνεργασίας μας με την Επιτροπή σας κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Οι σχέσεις ε, του ελεγκτικού συνεδρίου με την Επιτροπή σας είναι πάρα πολύ σημαντικές για να μπορέσει να υλοποιεί τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που τις εκχωρεί η συνθήκη, να επικουρεί δηλαδή το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο μάλλον στον έλεγχο και στη διαχείριση του προπολογισμού και να προάγει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία τα τελευταία τρία χρόνια έχει αρχίσει μια διαδικασία εσωτερικής μεταρρύθμισης στο Ελεκτικό συνέδριο με αυτοξιολόγηση και ε, ε, γενικότερο πλαίσιο διαχείρισης. Ε, εκπονήσαμε μια στρατηγική 2009-2012 για να βελτιωθούν να εντοπιστούν καλύτερα οι βελτιώσεις που χρειάζονται στους αντίστοιχους τομείς. Πολλές από τις ε, δράσεις προτεραιότητας που συνδέονται με τη στρατηγική αυτή έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Ε, μεταξύ αυτών και ε, η μεταρρύθμιση του εσωτερικού κανονισμού μας, όπως προβλέπεται από τη συνθήκη. Οι υπόλοιπες δράσεις θα υλοποιηθούν το 2011 και το 2012. Ωστόσο, οι δράσεις αυτές δεν αρκούν από μόνες τους για να εγγυηθούν ότι θα έχουμε τον στόχο και τον αντίκτυπο που επιθυμούμε χρειάζεται εμπιστοσύνη συνεχής ε, όλων των ενεχομένων φορέων και της δικής της Επιτροπής. Ε, σε θέματα εμπιστοσύνης, διαφάνεια και ε, η ανοιχτή συνεννόηση είναι απολύτως απαραίτητες. Είμαστε προσιλωμένοι στην ανεξαρτησία, στην ακαιρεότητα και ε, στην αμεροληψία του θεσμικού μας οργάνου. Ο επαγγελματισμό είναι πολύ σημαντικός και ε, η προστιθέμενη αξία που δημιουργείται ε, μετά από τη λειτουργία μας που βασίζεται πάντα στην αριστεία και στην αποτελεσματικότητα των συνεργατών μας. Σε αυτά τα στοιχεία οφείλουμε τη φήμη που χαίρει το θεσμικό μας όργανο τα τελευταία χρόνια και την εμπιστοσύνη μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Οι στόχοι της στρατηγικής για το 2009 2012 υλοποιούνται όπως σας είπα και θα ε, συνεχίσουν να καθοδηγούν το έργο μας και για το 2011. Η ανεξαρτησία, η κεραιότητα και η μεροληψία είναι βεβαίω απαραίτητα προαπαιτούμενα για οποιαδήποτε ε, αρχή ελέγχου και μάλιστα υψηλού επίπεδου. Ε, το, η συνθήκη μας ε, δίνει κάποια στοιχεία, κάποιες αρμοδιότητες μας, ε, στα θεσμικό όργανο και ε, ορίζονται και διαδικασίες για τον ορισμό των μελών. Ωστόσο όλες αυτές οι ρυθμίσεις και οι πρόνοιες από μόνους τους δεν αρκούν για να δημιουργηθούν εμπιστοσύνη. δημιουργηθεί εμπιστοσύνη. Χρειάζονται και άλλα τα μέλη και το προσωπικό θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε υψηλά ε, δεοντολογικά στάνταρ και στην εργασία τους και στις μεταξύ τους σχέσεις για να ε, παραμένει υψηλή η λειτουργία του οργάνου και αμερόληπτη. Αυτό θα συνεχιστεί στο 2011 όπως και στο παρελθόν ισχύει. Δεύτερον, το Ελεκτικό συνέδριο θα πρέπει να συνεχίζει να δηλώνει τα ευρήματά του με τρόπο ε, ισόρροπο. Ούτε να υπερβάλλει τα προβλήματα, ούτε να τα υποτιμά και να τα υποπαρουσιάζει, να τα παρουσιάζει πάντα δε στο σωστό τους πλαίσιο. Για να φτάσουμε σε αυτό, ε, κάνουμε ακροάσεις ε, πριν δημοσιεύουμε τα ευρήματά μας, πάντα τα ελέγχουμε με εσωτερικές διαδικασίες επαλήθευσης και συζητούνται εις βάθος από τα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου. Για να ξηθεί και να ανταποκριθεί στη φήμη του το ελεκτικό συνέδριο θα πρέπει να αναγνωρίζεται και ως υπόλογο το ίδιο και ως διαφανή στη λειτουργία του. Για το λόγο αυτό η διαδικασία απαλλαγή για το συνέδριο που συζητήσατε σήμερα το πρωί είναι τόσο σημαντική και γι' αυτό τη λαμβάνω και τόσο σοβαρά υπόψη. Για το λόγο αυτό, για παράδειγμα, ε, αναθέτουμε σε ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή να επαληθεύει ε, τους λογαριασμούς μας και τα ευρήματα και τα αποτελέσματά μας. Έχουμε δείκτες επίσης ε, που μετρούν τη δραστηριότητά μας και για πρώτη φορά φέτος συμπεριλαμβάνουμε και δείκτες που συνδέονται ε, με την ικανοποίηση των πελατών μας. Εμπειρογνώμονες ελεγκτές από υψηλού ε, επίπεδου ε, ελεγκτικές αρχές ε, μας ελέγχουν και μας το λεγόμενο peer review στην αξιολόγηση μεταξύ ίσων και στο μέλλον θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και για το 2011 όπως προβλέπεται στη στρατηγική μας για την περίοδο αυτή 2009-2012 δεσμευόμαστε στους ελέγχους αυτούς όχι μόνο για την ε, λογοδοσία μας αλλά για να βελτιωνόμαστε συνεχώς και δείχνουμε εκεί πόσο ε, επαγγελματίες είμαστε. Το ελεκτικό συνέδριο είναι προσιλωμένο στην προσπάθεια αυτή, χρησιμοποιεί τις υψηλότερες ισχύουσες προδιαγραφές και είναι στην πρώτη γραμμή ε, της διοίκησης και του ελέγχου. Το 2011 ε, θα εφαρμόσουμε τις νέες ε, προδιαγραφές που ισχύουν διεθνώς και εγκρίθηκαν το 2010 από τις αντίστοιχες αρχές. Συνεισφέραμε σημαντικά στην εκπόνηση πολλών τέτοιων στάνταρτς και συμμετείχαμε ενεργά στις αντίστοιχες ομάδες εργασίας αυτών των διεθνών οργανισμών ε, ανώτατων ελεγκτικών αρχών. Το 2011 θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με άλλες τέτοιες αρχές για μεγαλύτερη καινοτομία και περισσότερη εναρμόνιση στην προσέγγιση ε, στον έλεγχο των κοινοτικών κονδυλίων και ε, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τις ελεγκτικές τους αρχές. Κύριε Πρόεδρε, κατά την επιλογή και την υλοποίηση των εργασιών μας για το 2011, βασικό μας μέλημα ήταν να φέρουμε ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτό σημαίνει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί εκ των προτέρων. Το 2011 προβλέπουμε να δημοσιεύσουμε 45 ετήσιες εκθέσεις και για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης και ε, Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και άλλα όργανα. Η βασικότερη αποστολή μας ε, είναι ε, ο εσωτερικός έλεγχος του κοινοτικού προϋπολογισμού, η δήλωση αξιοπιστίας δηλαδή που βασίζεται ε, στην ετήσια έκθεση, στην οποία μάλλον βασίζεται η ετήσια έκθεση. Αυτό δείχνει τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι δαπάνες, ο προπολογισμό, συλλέγονται τα έσοδα, δεν γνωρίζετε αυτά έχουμε και μια ε, δεξαμενή σκέψη, ένα think tank, με επιρογνώμονες και εσωτερικούς δικούς μας ε, για να δούμε πώς μπορούμε περαιτέρω να βελτιώσουμε τον οικονομικό έλεγχο του Γενικού Προϋπολογισμού της Ένωσης. Αποφασίσαμε λοιπόν να επανακαθορίσουμε το πεδίο εφαρμογή ετήσια έκθεση για την εκτέλεση του προπολογισμού. Πρώτον, η ετήσια έκθεση για τον προπολογισμό του 2010 θα συμπεριλαμβάνει νέα αξιολόγηση με τίτλο Έρευνα και εσωτερικέ πολιτικέ που θα καλύπτει τι δαπάνε σε θέματα ερεύνη και άλλων εσωτερικών πολιτικών που στην αρχή και προηγουμένω ε, ε, ε, ενέπιπταν σε άλλε κατηγορίε. Επίσης, για το 2012 θα έχουμε ξεχωριστές εκθέσεις και κεφάλαια που θα αφιερώνονται στην ε, γεωργία και στην ανάπτυξη της υπαίθρου αλλά και στην περιφερειακή πολιτική ενέργεια και μεταφορές και ε, απασχόληση και κοινωνικά θέματα Εξωτερική βοήθεια, αναπτυξιακή βοήθεια, διεύρυνση, διοικητικέ δαπάνες και έσοδα επίσης θα καλυφθούν ε, όπως και στο παρελθόν θα παραμείνουν χωρίς αλλαγή. Θα πρέπει να εντοπίζουμε τις ανάγκες ε, των ενδιαφερομένων ε, και των ε, αποδεκτών των εκθέσεών μας συμπεριλαμβανομένης και της Επιτροπής στα διάφορα τμήματα, στους διάφορους τομείς για να περιορίσουμε τις ανισορροπίες και τις ασυμμετρίες. Βεβαίως θα λαμβάνονται πάντα υπόψη τα θέματα αποτελεσματικότητας καθώς και οικονομική οικονομικοί περιορισμοί. Για το 2010 ε, έχουμε ε, ε, εκθέσεις και για τις δραστηριότητες και τα πεπραγμένα των Γενικών Διευθυντών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, το ελεγκτικό συνέδριο διερευνά τον τρόπο να έχουμε προσθέμενη αξία με εθνικές αρχές ελέγχου, ε, με πιλωτικά προγράμματα, με εθνικά ελεγκτικά συνέδρια, ε, πιλωτικό πρόγραμμα στην Τσεχική Δημοκρατία και στις κάτω χώρες, ε, σε ό,τι αφορά τι γεωργικές δαπάνε. Αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα ε, θα ολοκληρωθεί φέτο και ε, θα αξιολογηθεί ω εμπειρία. Σε ό,τι αφορά τι δυτικέ δαπάνε των θεσμικών οργάνων, η ετήσια έκθεση για τον προπολογισμό του 2010 θα καταθέσει τα αποτελέσματα των ελέγχων εποπτείας όλων των θεσμικών οργάνων συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου. Το 2011 το Ελεκτικό Συνέδριο επίση θα ελέγξει τι επιπτώσεις ε, έχει η έκθεσή του στη λειτουργία της εξωτερικής υπηρεσίας, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης δηλαδή. Καθώς αυξάνονται οι αρμοδιότητες και ανάγκες, ε, αυξάνεται και η πίεση στο ελεκτικό συνέδριο και στους πόρους μας. Ε, στο νέο δημοσιονομικό κανονισμό που προτείνεται λοιπόν, προτείνουμε εμείς να αναθεωρηθεί και η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπορέσει το ελεγκτικό συνέδριο στο μέλλον να ασκεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εντολή του. αυτή τη στιγμή ολοκληρώσει ε, όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό του το ελεγκτικό συνέδριο ε, θα πρέπει να αρχίσει η εκπόνηση ειδικών εκθέσεων. Αυτές οι εκθέσεις και οι έλεγχοι μας επιτρέπουν πραγματικά να προτείνουμε ε, συγκεκριμένα σημεία με προστιθέμενη αξία με ιδιαίτερη σημασία για τους ενδιαφερομένους και θα μπορέσει έτσι το ελεκτικό συνέδριο να αναφέρεται στην ποιότητα των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα εργασίας μας είναι κατάλογο θεμάτων που προτίθεται το συνέδριο να εκδώσει ειδικέ εκθέσεις και να κάνει ε, έλεγχο το 2011. Σε ό,τι αφορά ε, το νέο μέσο πολιτικής γειτονίας και συνοχής το Ιανουάριο του 2011 ε, μια ειδική τέτοια έκθεση δημοσιεύτηκε για τον Νότιο Κάφκασο. Ε, προβλέπουμε τρεις νέες τέτοιες εκθέσεις για ε, θέματα και Ασίας και Λατινικής Αμερικής, ένα δεύτερο για την αναπτυξιακή βοήθεια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως για τη βασική εκπαίδευση στην υποσαχάρη Αφρική και η διαχείριση ε, των συστημάτων ε, κτηνιατρικών ελέγχων για εισαγωγές κρέατος. Κατά το υπόλοιπο του έτους ε, προτίθεται να δημοσιεύσει το ελεκτικό συνέδριο και άλλες ειδικέ εκθέσεις για τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013 ε, για τη ε, χρηματοοικονομική μηχανική, για τα μικροδάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το σύστημα ενιαίων πληρωμών, καθώς επίσης και μια συνέχεια στην ειδική έκθεση ε, και τη διαχείριση της Όλαφ. Το 2011 επίσης θα αρχίσουμε μια σειρά δράσεων για διάφορα θέματα και μεταξύ αυτών έλεγχος ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού ε, Κοινωνικού Ταμείου το 2006 και επίσης ε, για τις βασικές υγειονομικές προβλέψεις και το πόσιμο νερό στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα υπόλοιπα θα τα βρείτε στο έγγραφο που έχει δημοσιευθεί και στα βαρτήματα. Σας έχουν διαβιβαστεί αυτά. Επιπλέον, το ελεγκτικό συνέδριο ε, δημοσιεύει και γνωμοδοτήσεις. Αυτές ε, είτε κατόπιν ετήσεων των ε, θεσμικών οργάνων για κάποιες επιπτώσεις δημοσιονομικές, οικονομικές ε, των νομοθεσιών ή ως γενική συνεισφορά για την ε, διαχείριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2011 θα έχουμε πολλές νομοθετικές προτάσεις και αποφάσεις που θα έχουν ε, σημαντική επίπτωση στην οικονομική διαχείριση της Ένωσης τα επόμενα έτη. Πρώτον, ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός με τις εκτελεστικές του διατάξεις και ο κανονισμός για τους οργανισμούς, agencies. Επίσης, ε, το θέμα των ιδίων πόρων και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2013 και οι προτάσεις για ε, κλαδική τομεακή ρύθμιση των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνέδριο ε, χαιρετίζει τη δυνατότητα να βοηθήσει τις σκέψεις και τον προβληματισμό της δικής σας Επιτροπής προσβλέπω στην ανταλλαγή απόψεων τον Απρίλιο για τη ε, γνώμη του συνεδρίου για τους κινδύνους και τις ευκαιρίες στον προπολογισμό της Ένωσης και την πρόταση για τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό. Βεβαίως, τα μέλη μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουν για οτιδήποτε χρειάζεται. Επιπλέον, θα Έχουμε και νέες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, οικονομική διακυβέρνηση ως απόκριση στην οικονομική κρίση. Θα παρακολουθήσει στενά το Ελεκτικό συνέδριο και τις εξελίξεις αυτές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον ε, λογιστικό έλεγχο, ε, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια σε οποιοδήποτε μόνιμο μηχανισμό σταθερότητας. Το πρόγραμμα λοιπόν για το 2011 είναι πολύ φιλόδοξο. Η δυνατότητα τα μας να ανταποκριθούμε θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό στην προσήλωσή μας, στην πάγια ε, προσήλωση ε, στην αριστεία, στις ικανότητες, στα προσόντα των μελών μας. Διατηρούμε τις προσπάθειές μας να προσλαμβάνουμε τους σωστούς υπαλλήλους και να καλύπτουμε τις ε, θέσεις που χειρεύουν. Υποστηρίζουμε και τη σταδιοδρομία και την επαγγελματική κατάρτιση των υπαλλήλων καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας τους. Επιπλέον, Θέλουμε όλο και περισσότερο να προοδεύουμε ε, στην ισορροπία φίλους ε, όλα ε, τα τμήματα και σε όλα τα επίπεδα της διοίκησής μας. Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητά μας θα συνεχίσουμε και στη στρατηγική 2009-2012 να εφαρμόζουμε τους στόχους μας αξιοποιώντα καλύτερα τους πόρους μας και μεταξύ αυτών για έλεγχο λογιστικού, έλεγχο για τη δήλωση αξιοπιστίας και για τη βελτίωση των μεθόδων διαχείρισης. Το 2011 επίσης θα αρχίσουμε να βλέπουμε καρπούς ε, της προηγούμενης προσπάθειας μας ε, για το streamline στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Ε, πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι σχέσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου με την Επιτροπή σας είναι εκ των όνων για να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη και να είναι καλή συνεργασία στην Ένωση και να το βλέπουν αυτό και οι πολίτες ότι τα χρήματά τους πιάνουν τόπο έχουμε κοινούς στόχους, κοινέ προκλήσεις ε, και τα δύο όργανα. Συνεργαζόμενοι και πάλι το 2011 όπως και στο παρελθόν, Είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε κύριε Πρόεδρε να συνεισφέρουμε, να οικοδομήσουμε στα όσα ήδη έχουμε πετύχει ε, προς ε, επιπλέον μεγαλύτερο όφελος του Ευρωπαίου πολίτη στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαστε και εμείς πεπισμένοι ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων μας είναι ε, ουσιαστικότατη και προς όφελος ε, της Ένωσης και των πολιτών. Αν δεν έχετε παρατηρήσει για τα όσα μας είπε ο Πρόεδρος, α, έχουμε παρατηρήσεις, αλλιώς θα περνούσαμε στο επόμενο θέμα. Ο κύριος Μίλντερ. Μια πολύ εντυπωσιακή ομιλία. Νομίζω θα πρέπει να αντιδράσουμε. Το πρόγραμμα του ελεκτικού συνεδρίου είναι πράγματι πολύ φιλόδοξο. Έχω κοιτάξει τις μελέτες και τους ελέγχους που θα αναλυθούν και είναι πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω. Κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι οι μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές, αλλά όλοι μιλάνε για συνεργασίες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και αυτό σημαίνει περαιτέρω συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα διερευνήσετε είναι η διευκόλυνση εγγύησεων των μικρομεσαίων ε, επιχειρήσεων. Ε, η ερώτηση προς τον κύριο Καλτέρα είναι υπάρχει οποιαδήποτε πρόσφατη μελέτη ή δημοσίευση του ελεκτικού συνεδρίου σχετικά με τις συνεργασίες ε, ιδιωτικού δημόσιου τομέα όπως έχουν διεξαχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν γνωρίζω καθόλου, αλλά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι μέρος ε, ε, είναι, μέσα, είναι ένα, ένα όργανο το οποίο και το ελεκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκάγερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε Καλτέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ να μας παρουσιάσετε το πρόγραμμα εργασίας σας και είστε και στη διάθεση μας στη συζήτηση. Ευχαριστώ που ήρθατε στις Βρυξέλλες σήμερα το πρωί. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εξ ονόματος της δικής μου πολιτικής ομάδας και να σας συγχαρώ για την ανανέωση της θητείας σας, για τη δεύτερη θητεία. Συμπροματικά θα είχα δύο-τρεις ερωτήσεις για το πρόγραμμα εργασίας του 2011. Είναι εντυπωσιακό ο κατάλογος των μελετών που μας δώσατε. Τον είδα. Ε, για το τι προτίθεστε να δημοσιεύσετε ως συνέδριο το 2011 και χαίρομαι για τη συνεχιζόμενη συνεργασία μας. Είναι πολλά ενδιαφέροντα σημεία. Είχα την ευκαιρία να δω λίγο τις προμελέτες. Θα με ενδιαφέρε ε, να μάθω με βάση ποια κριτήρια επιλέγετε αυτές τις προκαταρκτικές μελέτες. Και μια δεύτερη ερώτηση που συνδέεται με την προηγούμενη λίγο. Ναι, εξής. Μήπως χρειάζεται προμελέτη η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που αναλαμβάνει τώρα. Ουσιαστικά ένα νέο θεσμικό όργανο. Με ένα ξεχωριστό χαρακτήρα. Γιατί ε, η επικεφαλής ταυτόχρονα είναι και μέλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ύπατη εκπρόσωπος Συμβουλίου. Τους περασμένους μήνες εργαστήκαμε πάρα πολύ σκληρά για να δώσουμε δημοσιονομικό κανονισμό σε αυτό το νέο όργανο και κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης για τους υπαλλήλους του. Και νομίζω ότι θα άξιζε τον κόπο πολύ νωρίς να κοιτάξουμε αν αυτά που επινοήσαμε για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης είναι τα σωστά. Με τη σωστή ε, διαχείριση. Ε, Τρίτον, ε, μιλήσατε για τη συνεδρίαση του Απριλίου. Θα το θεωρούσα χρήσιμο να την προγραμματίσουμε έτσι. αν δεν ξέρω, μήπως έχει ήδη προβλεφθεί η ημερομηνία. Ε, πάντως να μας απασχολήσει τότε το θέμα της έκθεσής μας για την απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι ε, συμπεράσματα θα έχετε συναγάγει ως τότε να το συζητήσουμε αυτό για την απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διευρευνήσουμε τη δυνατότητα συνεργασίας σε κάποια θέματα που ίσως να χωλένουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μακοβέη. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ ε, τον Πρόεδρο για την παρουσίασή του. Θα ήθελα να συζητήσουμε σε αυτή την Επιτροπή τα θέματα τα οποία έφεξε ο κ. Γκουίρτα στη συνέντευξή του και να τα εξετάσουμε. Η πρώτη ερώτηση είναι η εξή. Στην συνέντευξη ο κύριος Σκουίρτα δήλωσε και παραθέτω «Ήμουνα μια μοναδική φωνή στην έρημο» εξέταση του 2008 αναφέρει ότι θα πρέπει το προσωπικό να αναφέρει οποιαδήποτε απειλή στην εξαρτησία του. Αλλά καμία διαδικασία του ελεκτικού συνεδρίου δεν αναφέρεται σε οποιασδήποτε διαδικασίες που προβλέπονται πότε ε, θα εξετάσετε αυτή την κρίσιμη αδυναμία που υπάρχει. Δεύτερη ερώτηση. Ο κ. Αγκουίρντα επίση αναφέρθηκε στην παρουσίαση των αδυνατότερων αδελφών εντό του ελεκτικού συνεδρίου παραθέτω. Μερικά από αυτά τα ε, μέλη βρίσκονται ακόμα στι θέσει του. Θα εφαρμόσετε το άρθρο 4 παράγραφο 1 του κανονισμού που θεσπιστήκε το 2010 και τρίτη ερώτηση έχετε δεσμευτεί να υλοποιήσετε τις συστάσεις ε, εξέτασης ε, peer review στη στρατηγική. Ε, τώρα είμαστε στα μέσα της διαδικασίας. Ποια μέτρα έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής. Θα κάνετε μια ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης που να αφορά την τρέχουσα κατάσταση της στρατηγικής υλοποίησης. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πριν δώσω το λόγο σε άλλο συνάδελφο, να επενθυμίσω στη συνάδελφο Μακοβέη που ίσως απουσίαζε πριν, ότι στη συνεδρίαση των συντονιστών εξετάσαμε ήδη αυτό το ακαθόδες θέμα που εκ νέου αναφέρατε εσείς και τις επόμενες μέρες σε αυτή την Επιτροπή θα διεξαχθεί ξεχωριστή ακρόαση και του Πρόεδρου Καλτέρα και του πρώην μέλους του Ελεκτικού Συνεδρίου για να εξετάσουμε ε, αυτό το θέμα, το σοβαρό το θέμα της συνεντεύξεως. Ε, λοιπόν, ε, το έχουμε, έχουμε επιληφθεί το θέμα, το γνωρίζουμε. Κυρία Γιάλα Σέντερ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Καλδέιρα, το Πρόεδρο, για το πρόγραμμα εργασίας, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, υπάρχουν στοιχεία που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και που εμβαθύνουν στην ανάγκη που έχουμε για να κάνουμε τον έλεγχο και την παρακολούθηση του κοινοτικού προϋπολογισμού. Θα ήθελα να το, γνωρίσω, να το ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Για μια πρόταση γνωμοδότηση σε σχέση με τα στοιχεία για το ΑΕΠ που χρησιμοποιούνται Και όταν θα φτάσουμε και στη συζήτηση για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές. για τη στρατηγική αντιμετώπιση χρηματοοικονομικής κρίσης. Γιατί αυτή τη συγκεκριμένη νομοδότηση, σε τι αποσκοπείτε, τι θέλετε να διευκρινίσετε. Και στις προκατακτικές μελέτες βλέπουμε μία ε, που έχει να κάνει με τη διαχείριση της κρίσης και τα μέτρα που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενικά στο ευρωπαϊκό το χρηματοοικονομικό σύστημα και οικοδόμημα. Ποιοι είναι οι στόχοι ε, στους οποίους αποσκοπεί ε, το ελεκτικό συνέδριο. Γιατί θέλετε αυτή την προκατακτική μελέτη, γιατί θα έχει πολύ σημαντική επίπτωση και θετική εννοώ στις δημοσιονομικές προοπτικές της Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Καλτέρα για την παρουσίασή του και για την εξωτερική συνεργασία και θα ήθελα να τον συγχαρώ για την ε, έναξη της δεύτερης θητείας του. Σχετικά με τις δραστηριότητες του Ελεκτικού Συνεδρίου έχω μία ερώτηση. Συνήθως ε, κάνουμε πολύ πρακτικής φύσεως συζητήσεις και φαίνεται ότι το ελεκτικό συνέδριο δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό διότι έχουμε μόνο ένα μέλος αν κάτω μέλος και θα πίστευε κανείς ότι αυτό είναι αρκετά αποδοτικό αλλά έχετε αρκετή δουλειά για το κάθε μέλος του συνεδρίου ή μήπως θα πρέπει να το δούμε αυτό το σύστημα όπου το κάθε ε, μέλος έχει ένα έχει ένα Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι πάντα όταν σας βλέπω εδώ και χαιρόμαστε για τη συνέχιση της μελλοντική συνεργασίας. Πρέπει να πω στους συναδέλφους ότι στα πλαίσια για την έκθεση για την απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εργαστήκαμε εξαιρετικά και εντατικότατα. Ε, συνεργαστήκαμε πολύ. Θέλω να αναφερθώ σε μία πτυχή αυτή τη συνεργασία. Τα ξέρουν οι συνάδελφοι, το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα. Αλλά να το θέσουμε στο νέο πλαίσιο. Πρόκειται για τη λεγόμενη έκθεση αξιολόγησης που για πρώτη φορά ε, θα γίνει για το 2010 βάσει της τη Λισαβόνα. Αυτή η έκθεση απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον να μην μετράμε μόνο και να πρέπει να αποδεικνύουμε την νομιμότητα και την ορθότητα και την κανονικότητα αλλά και τη σκοπιμότητα στο μέλλον για τα πόσο είναι ε, σκόπιμα αυτά τα προγράμματα, κατά πόσο πιάνουν τόπο τα χρήματα. Θα πρέπει λοιπόν να μας ε, υποβληθεί αυτή η έκθεση. Και στις επαφές που είχαμε μαζί σας κύριε Καλτέρα συζητήσαμε για το ρόλο του δικού σας θεσμικού οργάνου. Δεν μπορώ να φανταστώ κανένα καλύτερο θεσμικό όργανο που να ταιριάζει να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, τουλάχιστον με τις ειδικέ έκτακτες εκθέσεις σας που πολλές φορές δεν αφορούν μόνο ε, τη, το νομότυπο, αλλά το σκόπιμο της κάθε δράσης. Ήδη από τώρα το κάνετε αυτό. Τώρα όμως είναι υποχρεωτικό. Ε, ob Sie diese Rolle wahrnehmen. Και θέλω να σας ε, ρωτήσω, ε, θα τον αναλάβετε αυτό το ρόλο, θα το υλοποιήσετε αυτό. Πήραμε ένα κατάλογο σήμερα στα αγγλικά, αλλά στον κατάλογο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απαλλαγή ε, γράφουμε κάπου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ορίσει ένα ειδικό εκπρόσωπο που να ασχολείται με τον ε, λογιστικό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των, δραστηριοτήτων της πάντα από αυτό το πρίσμα της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της σκοπιμότητας. Performance το λένε και Εσείς είστε πρόθυμοι να ε, αποτελέσετε ένα συνομιλητή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το λόγο κύριε Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Τα καλά λόγια απευθύνονται και σε μένα και στο ελεκτικό συνέδριο προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις τεθήσεις ερωτήσεις. Όσον αφορά αυτά που είπε ο κύριος Μούλτερ για το έργο του ελεκτικού συνεδρίου στα πλαίσια της συνεργασίας ιδιωτικού δημοσίου τομέα. Κάθε χρόνο να σας πω ότι ασχολούμαστε με αυτή τη συνεργασία που λαμβάνει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες τις κοινοπραξίες τις ελέγχουμε κάθε χρόνο και από τη φύση τους ε, είναι συνεργασία ιδιωτικού ε, δημόσια τομέα οπότε γίνεται ο έλεγχος αυτών των κοινοπραξιών. Ε, ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός προτείνει αντιμετώπιση του θέματος πιο διαρθρωμένα. Και όσον αφορά τον ίδιο συνομικό κανονισμό, πρέπει να λαμβάνονται κάποια μέτρα προφύλαξης και θέλουμε να αξιολογήσουμε νέα μέσα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στον τομέα. Όσον αφορά τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όπως ξέρετε, προβλέπεται τη συνθήκη. Άρα έχει την δικαιοδοσία να ελέγχει όλου του πόρου του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού που διοχετεύονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Ε, και αυτό πραγματοποιείται είτε μέσω του ελέγχου των μέτρων που εφαρμόζονται μέσω εντολής, όπως η περίπτωση που αναφέρθηκε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και του, ε, του μέσου που προβλέπεται ή των μέσων οικονομικής διαχείρισης που συνάδουν με τα διευθυντικά ταμεία για να υποστηρίξουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προσβλέπουμε στην εξέταση και αναφορά σε αυτά τα δύο συγκεκριμένα θέματα κατά τη διάρκεια ενεστώτος έτους και, και θέλουμε να δούμε ποια θα είναι η εντολή του δικαστηρίου όσον αφορά τα νέα μέσα και αν διαφυλάσσονται τα δικαιώματά μας επαρκώς. Αυτό είναι το μήνυμα που αποστέλουμε για το νέο δημοσιονομικό κανονισμό, αλλά ε, μέχρι τον Απρίλιο που προβλέπεται να καταλήξουν σε κάποια τοποθέτηση έχουμε περιθώρια. Το πρόγραμμα είναι πράγματι φιλόδοξο, ίσως και υπερβολικά φιλόδοξο. Προσπαθούμε όμως να κάνουμε καλύτερη βέλτιστη χρήση των πόρων και αναφέρονται κάποια στοιχεία σε αυτό το πρόγραμμα εργασίας για να απαντήσω το κ. Κάερ και τα κριτήρια είναι βασικά τέσσερα είναι ο κίνδυνος η σχέση όσον αφορά τις οικονομικές συνέπειες η κάλυψη και ο αντίκτυπος και βάσει αυτών των κριτηρίων γίνεται αξιολόγηση των θεμάτων. Α, με ύψιστη προτεραιότητα, μεσαία προτεραιότητα, μικρή προτεραιότητα. Εφόσον έχω περιορισμένους πόρους, βάζουμε πρώτα στον κατάλογο τα υψίστη σημασία θέματα. Γι' αυτό επιλέγουμε κάποια θέματα βάσει προτεραιότητας. Λοιπόν, τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη. Τη σημασία. Ποια αιτήματα κάνει το Κοινοβούλιο για να δώσει απαλλαγή. Και το Ταμείο Αλληλεγγύη και τα άλλα για τη μετανάστευση είναι αυτά που θέλουμε να εξετάσουμε σαν προτεραιότητα, όπω προσπαθήσαμε να ασχοληθούμε με άλλα θέματα που θα μπορούσαν επίση να συμπεριληφθούν σε εκθέσει σχετικά με άλλα εργαλεία διαθέσιμα για τη ρύθμιση των θεμάτων. Η υπηρεσία εξωτερική δράση. Έχουμε γνωμοδοτήσει δύο φορές για την προτινόμενη αλλαγή του κανονισμού για το προσωπικό και του δημοσιονομικού κανονισμού που σχετίζονται με αυτή την υπηρεσία εξωτερική δράση. Έχουν υποβληθεί γνωμοδοτήσεις και ήταν χρήσιμα για το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όταν ετοίμαζαν τι σχετικέ προτάσει δεν υπάρχει πρώτερη διαβούλευση με το ελεκτικό συνέδριο. Αυτή είναι πολιτική απόφαση του Συμβουλίου. Αλλά σε αυτές τις νομοδοτήσεις το ελεκτικό συνέδριο εκφράζει τις απόψεις του σχετικά με θέματα διαχείρισης των νέων υπηρεσιών, της νέας υπηρεσίας μάλλον, εξωτερικής δράσης και πώς να γίνει ο πραγματικός έλεγχος ε, της νέας ενίας, του νέου σχεδίου που εφαρμόζεται και υλοποιείται. Το 2011 πώς θα επηρεάσει εργασίες μας η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Διότι είναι ιονή θεσμικό όργανο, ιονή θεσμός. Πρέπει να δούμε πώς η διαδικασία απαλλαγή επίσης μπορεί να εφαρμοστεί. Ένα είναι σίγουρο. Όλα τα οικονομικά, οικονομικής φύσης που χειρίζεται η εξωτερική υπηρεσία θα ελεγχθούν ε, από τον Συμβούλιο, αυτά που είναι από την αιγύδα του Συμβουλίου το 2010, τα στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση των επιχειρήσεων που καλύπτονται από την αρχή του προπολογισμού και τα χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καλυφθούν. Θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη η μελλοντική όλων αυτών και πώς θα μπορέσουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο να διασκεδάσουν τις ησυχίες του Κοινοβουλίου και να διευκολύνουμε καλύτερο έλεγχο, ορθολογικό έλεγχο τη νέα υπηρεσία συναθρίζοντας δύο στοιχεία. Δύο χρηματοδοτικές πηγές που χρησιμοποιούν για να εφαρμόζουν, υλοποιούν τις δράσεις τους. Ίσως αυτή θα είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα με αυτή την Επιτροπή στην ετήσια συνάντηση. Ε, μάλλον στη συνάντησή μας αυτή μπορούμε να αλλάξουμε ενδεχομένως απόψεις και να δούμε ε, πώς μπορούμε να καλύψουμε ανησυχίες σας. Προς, τις προς την κυρία Μαρκοφέη να πω ότι αναφέραμε κάποια στοιχεία του κυρίου Έγκβη, τη συνεντεύξεις του κυρίου Έγκβη. Δεν είδαμε τις δύο δηλώσεις μετά, δεν τις ε, λάβαμε, έτσι εξετάσαμε δελεχώς, που εκεί αναλύει το νόημα των δηλώσεων του. Να πω δύο πράγματα μόνο όσον αφορά τα θέματα της ανεξαρτησίας των ελεγκτικών φορέων. Αυτά που αναφέρονται και από την ε, εξέταση των ομοτήμων. Ε, εξετάζουμε τη σχετική σύσταση και νομίζω ότι όλοι οι ελεγκτικοί φορείς πολύ σύντομα θα πρέπει να προβούν σε δήλωση ανεξαρτησίας αλλά εφαρμόσω τον κανονισμό DAF για το θέμα των whistleblowers. Ε, και δεν θα πρέπει, θα, κάποιος αποκλίνει από, το, από τον κανονισμό του Κοινοβουλίου πρέπει να εφαρμόζονται ε, ε οι πειθαρχικέ ε, Ο κύριος Έγκβη και στο European Voice και στην Focus Ten ανέφερε κάποια πράγματα και εκείνο θα σας πει τι εννοούσε. Το ελεγκτικό συνέδριο, σύμφωνα με τους δικούς του κανόνες, πρέπει να ασχολείται με θέματα παραβιάσεως των συνθήκων όσον αφορά την συμπεριφορά. Διαβάστε τα τις του κ. Βίντε, είναι πολύ σαφής σε αυτά που λέει. Ουδέν περαιτέρω σχόλιο. Σε ανοιχτή συνεδρίαση με τα χαράς να αναφερθώ σε όλα αυτά τα θέματα. Βέβαια, σήμερα ασχολούμαστε με το πρόγραμμα ε, αναφέρομαι στο πρόγραμμα εργασία. Αναφέρθηκα στο πρόγραμμα εργασία του ελεκτικού συνεδρίου. Η κυρία Γιάλα Σέντερ ανέφερε δύο πράγματα. Ποιοι είναι οι στόχοι μα όσον αφορά το GNI και την χρηματοστατική κρίση. Όσον αφορά την χρηματοστική κρίση, παρακολουθούμε τον εποπτικό πλαίσιο εκ του σύνεγγης των τρίων νέων εποπτικών φορέων που συνέστησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βάσης Αποφάσεων του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Βλέπουμε πώς λειτουργεί και τα πόσο είναι σωστή απόφαση της Επιτροπής. Εάν καλύπτονται όλα τα αναγκαία σημεία. Όσον αφορά το GNI, πρέπει να δούμε πώς έχει συνταχθεί και ποια είναι η συγκρισιμότητα, αν υπάρχει αξιοπιστία και συγκρισιμότητα στοιχείων θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό όσον αφορά τους ιδίους πόρους. Αφορά μακροοικονομικά στοιχεία αυτό το θέμα και στατιστικά στοιχεία και για άλλους σκοπούς, κυρίως δημοσιονομική προπτική ή άλλους τομείς όπως για το κρατικό χρέος κάποιων κρατών μελών. Θα μπορούσε λοιπόν να αποτελέσει το δέον εργαλείο και σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ τον κύριο Ιταλά για την ερώτησή του. Φοβούμαι όμως ότι σύμφωνα με τη συνθήκη χρειαζόμαστε ένα μέλος κατά κράτος μέλος. Μόνη λύση, σύμφωνα με την άποψή μου, μέχρι ότου αλλάξει η συνθήκη μπορούμε να αποχωρήσουμε περισσότερο. Η συνθήκη είναι αυτή που είναι. Στο παρόν πλαίσιο, ένα μέλος κατά κάτω μέλος, 27 μέλη στο συνέδριο, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνογνωσία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σύμφωνα με τους πόρους που έχουμε. Κάναμε σημαντικό βήμα το 2010 για τους ίδιους πόρους. Έχουμε ε, σε εξυγχρονίσει, έχουν κάνει πιο κομψή διαδικασία. Έχουν γίνει σωστή κατανομή των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων. Έχουμε γίνει πιο αποτελεσματικοί από τη χρήση των πόρων, θα έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα και οι διαδικασίε μα θα είναι κομψότερε και πιο εύκαμπτε. Αν υπάρχει προθυμία πολιτική και τα κράτη-μέλη θέλουν να αλλάξουν τη συνθήκη, είναι πρόθυμο το συνέδριο να συμβάλλει και να συμμετάσχει στη συζήτηση και προβλέπω ότι βλέποντας τα αποτελέσματα των μέτρων που ελήφθησαν στα πλαίσια αυτής της κρίσης, τα νέα οικονομικά μέσα, τους μηχανισμούς πληρωμών, τα μέτρα σταθερότητας που ανακοινώθηκαν μετά το 2013, θα έχουμε πολλές συνέπειες για το δημόσιο έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να δούμε τι προβλέπεται σήμερα στη συνθήκη όσον αφορά τον εξωτερικό δημόσιο έλεγχο της Ευρωπαϊκή Ένωση και το σχετικό πλαίσιο και τους περιορισμού. Και αν είναι αποτελεσματικό το πλαίσιο ή μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τη σύνθεση όμως του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου μπορούμε να την αλλάξουμε. Βλέποντας ποιες είναι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι αυξάνεται ο συντονισμό των δημοσιονομικών, φορολογικών, πολιτικών, οικονομικών πολιτικών. Άρα χρειάζεται ολοκλήρωση όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική διαχείριση, σοφή χρήση, συνετή χρήση των χρημάτων, ευέλικτους κανόνες, ευέλικτες διαδικασίες. Αν έχει την ίδια εντολή το ελεκτικό συνέδριο, Εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να προβλέψουμε και τι θα μπορέσουμε να κάνουμε και στο μέλλον. Είμαστε πρόθυμοι. Η ουσία του προβλήματος σημαντικότερο από τη σύνθεση των μελών. Όμως, αν υπάρχει πολιτική βούληση να αλλάξει συνθήκη, βεβαίως θα αλλάξει συνθήκη και θα πρέπει να ε, προσαρμοστούν δεόντω οι θεσμοί. Πρώτα όμω, να ασχοληθούμε με την ουσία πρέπει. να λάβουμε υπόψη τι τρέχουσε εξελίξει τη Ευρωπαϊκή Ενώση που έχουν τεράστιε συνέπειε όσον αφορά την εντολή του εξωτερικού ελεγκτικού φορέα. Σύμφωνα την παρούσα συνθήκη, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Ανέφερε κάποια ο κ. Μούλτερ. Συνεργασία ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Και άλλα οικονομικά μέσα. Όπως το Ταμείο Σταθερότητας είναι κάτι διακυβερνητικό. Αν θέλετε να κάνει κάτι, το ελεκτικό συνέθριο τι να κάνουμε. ιδιωτικό ε, το, ε, ιδιωτικό ταμείο ελέγχει ιδιωτικό ταμείο στο Λουξεμβούργο που ελέγχεται από ιδιωτικό ελεγκτικό φορέα που διέπεται από τον Λουξεμβουριανό νόμο. Τελεία και παύλα. Τι να κάνουμε εμείς. Αυτά τα θέματα πρέπει να εξετάσουμε. Κατάλαβα το ερώτημα βεβαίως, βεβαίω. Αλλά ε, η συνθήκη είναι αυτή που είναι και θα πρέπει να κινηθούμε σε αυτά τα πλαίσια. Στο δεδομένο πλαίσιο θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους μας. Στα αυτά που είπε ο κ. Χατζημαρκάκης, το ερώτημά σας. Ασχολείται με αυτό το θέμα. Εξελίξει την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας και πώς ανταποκρίνεται το ελεγκτικό συνέδριο. Το ελεγκτικό συνέδριο μπορεί να πει ότι θέλουμε να δούμε συγκεκριμένα ποιο είναι το περιεχόμενο της έκθεσης αξιολόγησης. Και σε αυτά τα πλαίσια τι μπορεί να κάνει το συνέδριο αν η έκθεση Φερρυπίν αναφέρεται σε επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή ποια ήταν η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε διάφορες τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ποιες ήταν επιδόσεις, τότε ποιο είναι ο ρόλος, ποια είναι η θέση του, του ελεκτικού συνεδρίου, πώς μας συμβάλλουμε στη συζήτηση που υπογράμμισε ο κ. Χατζημαρκάκης. Ε, εγώ θα έλεγα, α δούμε ποια θα είναι η μορφή τη έκθεση ποιο θα είναι το περιεχόμενο και πώ μπορεί το ελεκτικό συνέδριο να παράσχει διαβεβαιώσει στα ελεκτικά στα θεσμικά όργανα κατά πόσο αυτά που αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αξιόπιστα. Αυτή είναι η συμβολή μας. Αλλά τώρα προδικάζω. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι πρέπει να συμπεριλαμβάνει αυτή η έκθεση. Αυτό αφορά και την απαλλαγή. Μπορούσε στην ετήσια έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου να το αναφέρουμε αυτό, να προσθέσουμε αξία με νέα κεφάλαια στα οποία εξετάζουμε τις επιδόσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής πόσο αποτελεσματική είναι η οικονομική διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης. Αυτά είναι θέματα χρονικού συντονισμού, ε, εκπώνηση εκθέσεως αξιολογήσεως, διαθεσιμότητας των πληροφοριών, έγκαιρη διάθεση των πληροφοριών. Ένα από τα προβλήματα που έχουμε είναι το χρονοδιάγραμμα για την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων που εκπονεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έρχεται πολύ αργά η έκθεση. Πολύ κοντά στην προθεσμία πρέπει εμεί να, να υποβάλουμε τη δική μα ε, έκθεση. Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αλλά θα δούμε ποιο καλύτερο δυνατό τρόπο μπορούμε να κινηθούμε για να βοηθήσουμε το θεσμικό αυτό όργανο, το Κοινοβούλιο, να αντιμετωπίσει τι νέε εξελίξει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τι απαντήσει σα. Ευχαριστούμε λοιπόν τον πρόεδρο Καλντέρα, τον οποίον αποχαιρετούμε και πάμε συνεδρίαση των συντονιστών και κλεισμένων των θερών. Θα παραμείνουν μόνο οι συντονιστές των διαφόρων πολιτικών ομάδων.